Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι 8 και 38. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Ας ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Πάμε στο σημείο υπαρήθω 8. Ε, χορήγηση εγγύηση Ευρωπαϊκή Ενώση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών και από χρηματοδοτικέ δραστηριότητε που υποστηρίζουν επενδυτικά ρεκτό εκτό τη Ένωση. Ο κ. Κούκαν είναι ο συντάκτης. Ε, έχει να πει κάτι. Δεν είναι καν εδώ, άρα τι να πει. Άρα πάμε αμέσω στη ψηφοφορία. Ωραία. Πού να ξεκινήσουμε. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές. Ας γίνει έλεγχος για τη 40. Ξεκινάμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη. 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε τι γίνεται με τη 49 Άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιος συνάδελφος δεν συμμετέχει πέρας και απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 26 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική ψηφοφορία του σχεδίου γνωμοδοτήσεως που τροποποιήθηκε. Άρχεται. Συμμετέχουν και 51, πέρας, εγκρίνεται με 39-8. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο σημείο. Ταμείο Εγγυήσεων για τις Εξωτερικές Δράσεις. Ο κύριος Κούκαν είναι ο συντάκτης. Πάμε αμέσως στην ψηφοφορία. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3, υπέρ. Α, ναι, ναι, ναι, συγγνώμη. Καταπίπτει. Ναι, ναι, εγκρίθηκε, ναι, έξι. Πάμε λοιπόν στην 8. Όχι, όχι. Καταπίπτει η 3, λέει ο πρόεδρος. Α, ωραία, εντάξει. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, 1 καταπίπτει, Ψηφίζουμε την 1. Μου λέγουν ότι πρέπει να ψηφίσουμε την 1. Υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε. 1. Άρχεται. Πέρας. 31-19. 5 υπέρ. όχι. Mm, καταπίπτει αυτή. Άρα ηλεκτρονική ψηφοφορία, η τελική, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 43 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά. Σημείο 10. Υπογραφή του πρωτοκόλλου τη Συμφωνία Πλαισίου Εταιρική Σχέσεω και Συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώση και των Κατών μελών τη αφενό και τη Μογγολία αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση τη Δημοκρατία τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εισηγητή ο Χέλμοντ Σόλτ. Θέλετε να πείτε κάτι, μήπω. Όχι. Οπότε ψηφίζουμε κατευθείαν. Πω, περίπλοκη ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία ξεκινάει. Πέρας. 49-1. Εγκρίνεται. Οπότε είμαστε ακριβώς στην ώρα μας. Και ερχόμαστε στο σημείο υπαριθμών 11. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Άνταμ Σουμπ επιτετραμένο της αποστολής των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άνταμ, θες να είσαι εδώ. Would you like your colleague to sit next to you? Uh, no, no, I think I'm okay. Uh, no. I think we're easy. Ladies Κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μου που καλωσορίζω τον Άνταμ Σουμπ, επιτετραμένο της αποστολής των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τις Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τις Πολιτείες Αμερικής. Πολλοί από εσά θα γνωρίζετε ότι ο κύριος Σουμπ είναι διπλωμάτης καριέρας, έφτασε το 2015 στις Βρυξέλλες και ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2017. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τις οποίες είχα την τιμή να προεδρεύω στο παρελθόν. Ο Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας τον είπα, είναι εδώ. Καλώς ήρθατε. Ε, πιστεύω ότι η πρωινή μας αυτή συνεδρίαση δείχνει ότι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι κοντά στους ε, πιο στενούς ε, συνεργάτε και συμμάχους. Ο πρόεδρος ο κ. Τρόμπα έστειλε ισχυρό μήνυμα όταν μίλησε στο Κογκρέσο, είπε ότι οι ΗΠΑ Πολιτείες και παραθέτω υποστηρίζουν ένθερμα τον ΝΑΤΟ, μια συμμαχία που ήταν ένα δεσμό μετά το δεύτερο, που δημιούργησε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που νίκησε το φασισμό και τον κομμουνισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ ποτέ δεν είχαν τόσο ισχυρή διατλαντική α, σχέση όσο τα προηγούμενα 2,5 χρόνια της κοινοβουλευτικής αυτής θητείας. Είναι πολύτιμη αυτή η σχέση, θέλουμε να συνεχιστεί, κυρίως στα πλαίσια των παρόντων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η διεθνής ε, κοινότης. Αγαπητέ Άνταμ Σουμπ, θέλω διαβεβαιώσεις από σας τα μέλη όσον αφορά τις διεθνείς δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ΗΠΑ σχετικά με το Ιράν Φερρυπίν και τις πολιτικές για την επίλυση της κρίσης στην Συρία, Λιβύα, Ιμένη και Ουκρανία, για να αναφέρω κάποια από τα προβλήματα. Προτείνω να δώσουμε στον κύριο Σούμπα το λόγο για ένα δεκάλεπτο πάνω κάτω και μετά να έχουμε αρκετό χρόνο για να έχουμε μια καλή και ελπίζω καρποφόρα συζήτηση. Καλώς ήρθατε, ένα θερμό καλωσόρισμα και έχετε το λόγο κύριε Σούμπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μακάλιστα συγχαρητήρια σε εσά και στου άλλου ευρωβουλευτέ για του νέου ηγετικού σα ε, ρόλου στην Επιτροπή. Μεγάλη χαρά για μένα και τιμή για μένα να απευθυνθώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα και να μοιραστώ τι απόψει ε, τη νέα Αμερικανική κυβερνήσεω, όσα γνωρίζουμε τη θέση τη και πώ βλέπετε εσεί τη διατρατική σχέση, πώ τη βλέπετε να εξελίσσεται του επόμενου ε, μήνε, όπω προανέφερα σε συναντήσει με αρκετού από εσά, σε αυτή την αίθουσα, το έργο των διπλωματών τη, τον είναι καταρχάς να προσπαθούμε να μεταφράζουμε τις απόψεις της ηγεσία μας στη Ουάσιγκτον για τους εταίρους μας στο εξωτερικό και να ενημερώνουμε και την ηγεσία μας για αυτά που ακούμε και να δίνουμε την καλύτερη δυνατή συμβουλή για να προωθούμε τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της μεταβάσεως. Η αποστολή μας, η αντιπροσωπεία μας των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προωθήσει τα καθήκοντά τη σοβαρά. Εξηγήσαμε στη νέα κυβέρνηση στη Ουάσιγκτον τη σημασία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή θεσμοί και την ε, αξία συνεχούς ισχυρής σχέσεως σύμπραξης Ευρωπαϊκής όπω είπα, σαν πυλώνα παγκόσμια ευημερίας, ειρηνή και σταθερότητα. Ελπίζω να είναι σημαντική γέφυρα την προσωπία μεταξύ Βρυξελών και Ουάσιγκτον και βλέπω ότι η σημερινή συνομιλία μα είναι μια μεγάλη δυνατότητα να το προωθήσουμε αυτό. Τον περασμένο μήνα είχαμε την ευτυχία να καλωσορίσουμε τον Αντιπρόεδρο Πεν ε, στις Βρυξέλλες ήθελε να συναντήσει μέλη ο κύριος Πέντ του Ευρωκοινοβουλίου αλλά ήσασταν στο Στρασβούργο σε συζητήσεις με τον Προέδρου Στούσκ Γιούνκερ και την είπατε εκπρόσωπη την κυρία Μογκερίνη και τις δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Πένς που θα ακούσατε ο Αντιπρόεδρος ο κύριος Πένς εξέφρασε τη δέσμευσή του Τη δέσμευση των ΗΠΑ για συνεχή συνεργασία και σύμπραξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση διαβίβασε τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για να είναι στο πλευρό της Ευρώπης, διότι δεσμευόμεθα από τις ίδιες εξέπαινες ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Και αυτή η δέσμευση δεν είναι πουθενά σαφέστερη από τα αντίστοιχα κοινοβούλια μα. Όπω γνωρίζετε, πολλοί από εσά, ίσω περισσότεροι από εσά, επισκέφτεστε συχνά τα μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ και είναι παρόμοιο το συνέστημα που επικρατεί στο Καπιτόλιο. Ε, είχα συνοδεύσει τον David με την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στη Ουάσιγκτον το Δεκέμβριο για τη διάλογο που έγινε στη Ουάσιγκτον και ήταν σαφέστατο για μένα και για του περισσότερου από εσά η κατάσταση στο συνέστημα. Θέλουμε υποστήριξη και από τι δύο πλευρέ τη διατρανική σχέση. Αυτό το βλέπουμε να ισχύει και στη Ουάσιγκτον. Θέλουμε τις σχέσεις με την Ευρώπη. πολύ στην Ευρώπη καλώς τα καθησυχητικά λόγια του Προέδρου του Αντιπροέδρου και άλλων οντά των αξιωματούχων των ΗΠΑ. Επίση ε, υπάρχουν όμω ε, και αρκετέ αβεβαιότητε, το καταλαβαίνω, όσον αφορά τη μελλοντική κατεύθυνση των πολιτικών που θα ακολουθηθούν. Αυτό αφορά εν μέρη και τη μετάβαση από μια κυβέρνηση σε άλλη. Ευτυχώ υπάρχουν βασικά μέλη ήδη τέσσερα. Έχουμε τον κύριο Τέλο, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Τζέφ Μάτι, Υπουργό Αμήνε, τον νέο σύμβουλο Μακμάστερ για θέματα εθνική ε, ασφαλεία αλλά πολλοί εργασιακέ θέσει πρέπει να καλυφθούν, κυρίω στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεύτερο και τρίτο επίπεδο αξιωματούχων και βέβαια νέο πρεσβευτή που θα στείλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η διαδικασία χρειάζεται χρόνο, αλλά εντωμεταξύ η πρόθεσή μου είναι να πλησιάσω στο το δυνατόν περισσότερο από εσά εδώ και στο Στρασβούργο σε μερικέ εβδομάδε, ούτω ώστε να οικοδομήσουμε στην βασική σχέση που έχουμε με τα, με τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ενώση σε μερικέ ημέρε θα συναντηθούν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενώσης στη Ρώμη για την, επέτειο, την 60η επέτειο της υπογραφής συνθήκης της Ρώμης. γιορτάζεται από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα, αύριο. Α, σήμερα το γιορτάζεται. Μεταξύ άλλων θεμάτων, οι ηγέτες παλεύουν με το πώς θα ανταποκριθούν στα επαιτήσει των ευρωπαϊκών ψηφοφόρων για την ασφάλεια στον γρήγορα μεταλλασσόμενο κόσμο και πώ θα διαχειριστούν τα αποτελέσματα τη παγκοσμιοποίηση. Είναι παρόμοια με τα θέματα που συζητούμε στη ΣΥΠΑ. Οι πολίτε ζητούν από του ηγέτε να δώσουν καλύτερη άμυνα κατά εξωτερικών απειλών. Χρειάζεται σωστή προσέγγιση στην καταπολέμηση τη δημοκρατία, αυστηρότερο έλεγχο των συνόρων και ε, ε, ε, ασφάλεια οικονομική αλλά και ακριβοδίκη. Αυτή η κοινή στόχη και από τι δύο πλευρέ του Ατλαντικού σημαίνει ότι έχουμε και ισοδύναμε ευκαιρίε για συνεργασία ίσες ευκαιρίες. Ακροθυγώς θα τα αναφέρω και θα ήθελα να ακούσω και σκέψεις πώς να βελτιωθεί η συνεργασία μας ε, και να έχουμε ένα θετικό θεματολόγιο από αυτόν. Λοιπόν, το πρώτα απ' όλα είναι άμυνα. Το πρώτο. Βασικός πυλώνας της λογικής άμυνας είναι το ΝΑΤΟ, η πιο επιτυχή στρατιωτική ε, συμμαχία στην ιστορία. Πρόσφατα, σε ανταπόκριση στην απειλή της Ρωσίας, βελτίωσε την εσωτερική θέση με τέσσερις μονάδες στην Πολωνία και στα Βαλτικά κράτη ε, για να έχουν μεγαλύτερη παρουσία και όταν ε, ο κ. Μάτη επισκέφθηκε το ΝΑΤΟ, τόνισε ότι οι δράσει τη Ρωσία παραβιάζουν το διεθνέ δίκαιο και αποσταθεροποιούν την όλη κατάσταση. Θα είμαστε αποφασιστικοί, θέλουμε να θαρρύνουμε του Ρώσου να συμμορφωθούν τι υποχρεώσει του στη συμφωνία του Μίνσκ, πλήρη εφαρμογή. Αυτή είναι προαπαιτούμενο για να αρθούν οι κυρώσει και αυτό δεν έχει αλλάξει. Ο Υπουργό κ. Τηλέσον ε, είπε ότι υποστηρίζει τη συμφωνία του Μίνσκ και θέλει να συνεργαστεί για να αποκλιμακωθεί η βία στην Ουκρανία. Και ο πρέσβη ο Νίκ Χέιλι, στο Ηνωμένο Εθνή, είπε ότι καταδικάζει τι δράσει στην Ουκρανία, τι ρωσικέ στην Ουκρανία, είπα. Και οι κυρώσει που αφορούσαν την Κρυμαία θα παραμείνουν μέσω όσου ε, ξαναδώσει την κυριαρχία τη Κρυμαία στην Ουκρανία. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, και δεν είναι η πρώτη, πιστεύει ότι η ειρήνη χρειάζεται ισχύ, ανταποκρίνηση ισχύ. Και θέλουμε να υποστηρίξουμε του συμμάχου στην Ευρώπη. Θα πρέπει όμω να μοιραστούμε τι ευθύνε μαζί τη διατλαντική ασφαλεία υπό το φως των δράσεων των Ρώσων. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει να, να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες ουσιαστικά. Καλωσορίζουμε την έκκληση του Συμβουλίου να, στα κάτι μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και την ανάγκη οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να πρέπει να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν το 2014, δηλαδή να αφιερώνουν το 2% του ΑΕΠΣ για τα αμυντικά. Θέλουμε να ενισχυθεί και άμυνα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πλαίσια παγκόσμια στρατηγική και πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Ευρωπαϊκή Νότο στη δήλωση τη Βαρσοβία θέλουν να αυξήσουν την αντοχή και άμυνα έναντι υβριδικών απειλών, άμυνα όσον αφορά τι απειλέ του κυβερνοχώρου και την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφόρων που εγγυηθούμε. Η αντικαταπολέμηση τη τρομοκρατία αυτή την εβδομάδα γίνεται διάσκεψη καταπολέμηση του ISIL. Δυστυχώ είδαμε κάποιε φρικτέ τρομοκρατικέ επιθέσει στις 22 είναι η επέτειος των τραγικών επιθέσεων στο σταθμό του Μάλμπεκ και του, που είναι κοντά εδώ και στο αεροδρόμιο των Βρυξελών. Πρέπει να συνεργαστούμε να αποφύγουμε κι άλλες τέτοιες επιθέσεις. Ε, λοιπόν, Θέλουμε να συζητήσουμε στο τελειό τη διαπολέμηση του ISIS ή ISIL, ε, συλλογικέ προσπάθειε στρατιωτικέ, να καταπολεμήσουμε του κρεσμαχητέ, να καταπολεμήσουμε την χρηματοδότηση των ε, τρομοκρατικών οργανώσεων και θα πρέπει ε, να βοηθήσει, έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργαζόμαστε στενά στην Ευρωπόλ, ανταλλάσσουμε εμπειρίε όσον αφορά τα ασφαλή σύνορα, ανταλλαγή πληροφοριών για να εξαλείψουμε τα ευάλωτα στοιχεία τη σε αυτό το τομέα προστασία τη ιδιωτικότητα, συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση είπα, DPPA, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε να μοιραζόμαστε πληροφορίε όσον αφορά τι δυνάμει τη τάξη, όσον αφορά τι ε, δραστηριότητε ε, των εγκληματικών ομάδων και των μοκρατών. Πρέπει να παραδεχτούμε επίση ότι το Ιράν εξακολουθεί να είναι ε, η χώρα που τονώνει και υποστηρίζει την τρομοκρατία και αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή, στη Συρία, στο Λίβανο και στην Ιεμένη. Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να εξασφαλίσουν ότι το Ιράν ποτέ δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο που θα μπορεί να απειλήσει είτε τις ΗΠΑ είτε του συμμάχους των ΗΠΑ. Να αναφέρω κάτι για τα σύνορα πάρα πολύ σύντομα και από τι δύο πλευρέ του Ατλαντικού οι ηγέτε προσπαθούν να, να βελτιώσουν τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και, και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη και να εξασφαλίσουν ότι εκείνοι που εισέρχονται δεν προτίθενται να βλάψουν. Λοιπόν, οι απειλέ για την ασφάλεια αλλάζουν και μεταλλάσσονται, οπότε η κοινή λογική δείχνει ότι συνεχώ θα πρέπει να επανεξετάζουμε και να αξιολογούμε τα συστήματα στα οποία βασιζόμαστε για να προστατεύουμε του πληθυσμού μα. Γνωρίζουμε τόσο τα βήματα που έκανε η κυβέρνηση μέσω ε, διαταγμάτων. Στοιχεία των διαταγμάτων αυτών ε, εξετάζονται δικαστικώ. Περιμένουμε να αποκριθούμε στι διεθνεί μα υποχρεώσει. Σεβασμό των ετούντων άσυλο και των προσφύγων ο Υπουργό ο κ. το σε αυτό τα ανθρώπινα δικαιώματα ακρογωνίω λίθο τη πολιτική των ΗΠΑ και θα έχουν επιφανή ρόλο και στο μέλλον όσον αφορά τη διαμόρφωση των πολιτικών μα. Συζήτηση, όπω γνωρίζετε, συνεχίζεται στην Ευρώπη. Ενίσχυση των μέσων και των, των φορέων όπω Σέγγεν, υπηρεσία πληροφοριών Σέγγεν, υπηρεσία για τι θεωρήσει Σέγγεν, Frontex κλπ. Τέλο, κάτι που με απασχολεί πολύ και νομίζω ότι απασχολεί κάθε πολίτη είναι η οικονομική ασφάλεια. Λοιπόν, τα ωφέλη της παγκοσμιοποίησης είναι προφανή σε όλους μας σε αυτή την αίθουσα, στη φυσαλίδα της Ουάσιγκτον, τη φυσαλίδα των Βρυξελών, σε τομείς που έχουν ωφεληθεί, αλλά υπάρχουν και πολλά μέρη σε όλες τις χώρες μας όπου οι πολίτες εκεί δεν έχουν ωφεληθεί από την παγκοσμιοποίηση και θα πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το κόστο και να εκτιμήσουμε το κόστο τη παγκοσμιοποίηση. Κάποιε ομάδε έχουν πληγεί σκληρότερα από άλλου στην κοινωνία και οι ηγέτε φέρουν ευθύνη να δημιουργήσουν συνθήκες όπου κάθε πολίτης έχει δυνατότητα να επιτύχει. Πουθενά δεν ήταν πιο ε, σοβαρή αυτή η συζήτηση από τον τομέα του εμπορίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει τολμηρό βήμα να επικυρώσει τη ΣΕΤΑ παρά την πολιτική αντίδραση που υπήρχε και θέλουμε να δούμε πώς η ευρωπαϊκή συζήτηση θα εξελιχθεί όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας και να δούμε τι στρατηγικές θα εφαρμόσετε ώστε να κατανοήσουν τα ωφέλη της συμφωνίας οι πολίτες. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιστεύει ότι ισχυρέ και δίκαιε συμφωνίε στον αφορά εμπόριο μπορούν να προωθήσουν την οικονομία, να δημιουργήσουν θέσει απασχόληση και να ζωγονήσουν τι κοινότητε που υποφέρουν. Η κυβέρνηση αξιολογεί τώρα το καθεστώς Ατλαντικών Συμφωνία, του TTIP, τη συμφωνία TTIP. Λοιπόν, γενικό στόχο εμπορική πολιτική είναι να επεκτείνουμε το εμπόριο με έναν τρόπο που είναι πιο ελεύθερο και πιο δίκαιο για του πολίτε. Για αυτή την κυβέρνηση αυτό δείχνει ότι πρέπει να έχουμε πιο αποτελεσματικά, αποτελεσματικούς θεσμούς που διέπουν το εμπόριο όπως ε, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Θα εξασφαλίσουμε ότι η ΕΠΑ που συμμορφώνεται με τις επιταγές του ΠΟΕ θα μπορεί να προωθήσει τα αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα, αλλά διαβεβαιώνουμε και ότι τα άλλα μέλη του ΠΟΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν πλήρω τι υποχρεώσει που έχουν αναλάβει. Πιο συγκεκριμένα συζήτηση για την οικονομία τη αγορά, το καθεστώ οικονομία τη αγορά τη Κίνα που συζητήθηκε εδώ και αλλού. Είναι ένα θέμα που συζητείται λοιπόν. Η συζήτησή μα δείχνει ότι έχουμε κοινά συμφέροντα και ευθύνε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλε οι χώρε συμμορφώνονται πλήρω με τι υποχρεώσει που έχουν αναλάβει στα πλαίσια του ΠΟΕ. Και πέρα από αυτό, το εμπόριο σε υπηρεσίε και αγαθά και σε επενδύσεις. Το εμπόριο αυτό. Πριν σταματήσουμε για ρωτήσει να επαναλάβω κάτι. Έχουμε ανάμεσα τη δέσμευση. Η χώρα μου στη διατλαντική σχέση θέλει να υποστηρίξει και το ευρωπαϊκό εγχείρημα και τι διατλαντικέ σχέσει. Αυτό και από τι δύο πλευρέ υποστηρίζεται και τα δύο κόμματα μάλλον και δύο πλευρέ από τον JFK ε, μέχρι τον Ρούνα Λίγκα υποστήριζαν την προσέγγιση. Είναι το μόνο θεσμικό όργανο που είναι άμεσα αιρετό ε, είναι το Ευρωκοινοβούλιο και στηρίζει αυτή τη σχέση. Και θα πρέπει η συνεργασία μα να είναι η βάση για την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι σημαντικό εταίρο για μα, όπω θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στι ανάγκε των πολιτών μα και να διαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση για του πολίτε μα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Άνταμ, για τις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση υπήρχε μεγάλη επιθυμία στην παρουσία Επιτροπή να ακούσουμε τα σχόλια του εκπροσώπου της το δυνατόν συντομότερο. Βλέπετε και από την λίστα των ονομάτων των συναδέλφων που εγγράφηκαν για να ζητήσουν το λόγο, τι μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει. Μία ώρα περίπου έχουμε χρόνο, δηλαδή μέχρι τις 10. Θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο σε όλους τους εγγεγραμμένους συναδέλφους. Πρώτα όμως θα ήθελα να δώσω το λόγο βεβαίως στην αντιπρόεδρο της ε, αντιπροσωπείας ε, για τις σχέσεις με τα αμερικάνικα νομοθετικά σώματα που εκπροσωπεί τον ε, πρόεδρο της αντιπροσωπείας κ. Έλε. Ζητώ συγγνώμη για την ε, ε απουσία του κ. Έλε, ο ίδιος ζητήσει συγγνώμη δηλαδή, έχω ορισμένα σχόλια μετά από τις παρατηρήσεις σας, οι οποίες συμφωνούν και με τα όσα διεπίστωσε το Προεδρείο μας όταν πήγαμε στην Ουάσιγκτον τον προηγούμενο μήνα. Και η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες ικανοποιούνται από τις παρατηρήσεις αυτές. Για πολλούς από εμά όμως ε, ανησυχούμε διότι ε, χρειάζονται διαβεβαιώσεις, διότι χρειάζονται ε, οι διαβεβαιώσεις αυτές. Έχουν πάρει μια τροπή οι σχέσεις μεταξύ των πλευρών που δεν αναμέναμε. Είπατε και εσείς ότι πολλοί ακόμα, πολλά πράγματα ακόμα είναι άγνωστα από την πλευρά της Ουάσιγκτον. Πάντως επιβεβαιώσαμε σταθερά ως αντιπροσωπεία ότι κάποιες παράλληλες μορφές πολιτικές με κάποιες στρατηγικές που προωθούσαν σύμβουλοι του Λευκού Οίκου θα είναι ανεπιθύμητες. Άκουσα με ικανοποίηση τα λόγια σας σχετικά με την δέσμευση υπέρ της κοινής ασφάλειας, υπέρ της συμμαχίας ΝΑΤΟ, υπέρ της συμφωνίας Μίνσκ σχετικά με τον ρόλο της Ρωσίας και την βία στην Ουκρανία. Θα ήθελα να ακούσω λίγα περισσότερα για τη Συρία. Μιλήσατε για τον ρόλο του Ιράν, αλλά να μην λησμονούμε ποιο είναι ο ρόλος του Κρεμλίνου στη Συρία. Εν τέλει θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για το εμπόριο. Η συνάντηση των G20 και η δήλωση ναύτα TPP, TPP, που νομίζετε ότι κατευθύνεται πραγματικά η κυβέρνηση Τραμπ και πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε να δούμε την κινέζικη κυβέρνηση να γράφει στα λάβαρά της την αποαγκοσμιοποίηση ενώ έχει βαθιές και θεμελιώδεις αλλαγές από τις δικές μας κοινέ αξίες. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να ενισχύσουμε ένα σύστημα βασισμένο σε αξίες, αλλά όχι μόνο σε συμφέροντα, σε βαθύτερες κοινέ αξίες. Νομίζω ότι υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος να δούμε ένα κόσμο που εν τέλει να μην ωφελεί ούτε τη μια ούτε την άλλη πλευρά. Ενώ αυτό που χρειάζεται είναι μια αμοιβαία υποφελή σχέση, η οποία έχει βαθύνει τι τελευταίε δεκαετίε και η οποία πρέπει να εξυπηρετεί και τι επερχόμενε γενναίε. Πρόεδρο Μακάλιστερ, ευχαριστώ κυρία Χάκεν. Προτείνω τώρα να ακούσουμε του συναδέλφου τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Α ε, περιοριστούμε όλοι σε δύο λεπτά το πολύ, διότι έχουμε πολλού που έχουν εγγραφεί. Και Άνταμ, όταν θα θεωρήσετε ότι φτάνουν οι ερωτήσεις για τον πρώτο γύρο, κάντε μας ένα σήμα για να μπορέσετε να απαντήσετε στον πρώτο γύρο των συναδέλφων. Την αντιπρόεδρό μας θα αρχίσουμε. Ευχαριστώ, ε, David. Ευχαριστώ τον κύριο Σουπ που ε, προσήλθε ενώπιόν μας. Μετέβην και εγώ με την αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου. Δεν γνωρίζαμε τίποτε ακόμη για την νέα κυβέρνηση, ήταν ένα είδος καινού χώρου. Τώρα βλέπουμε βέβαια κάποια ίχνη των πολιτικών που επιθυμεί να ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ για το πρώτο μέρος που μιλήσατε για την ασφάλεια και όπου είπατε ότι κοινό μας στόχος είναι η ασφάλεια και ότι οι διατλαντικές σχέσεις θα συνεχιστούν. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από τα όσα άκουσα για τη Συμφωνία Μίνσκ για την, κοινή, για την κινητή πολιτική ασφαλείας, για το ΝΑΤΟ. Όμως στο δεύτερο μέρος της δηλώσεώς σας, αυτό μου φάνηκε ότι δεν ήταν απόλυτα ξεκάθαρο. Θα ήθελα να διευκρινίσετε τις θέσεις σας, την πολιτική σας, για την συμφωνία TTIP. Έχουν διεξαχθεί 14 γύρι διαπραγματεύσεων και είχαμε φτάσει σχεδόν στο τέλος, στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αυτών. Μπορείτε να πείτε λίγα περισσότερα λοιπόν για τις εμπορικές συμφωνίες, για το μέλλον των εμπορικών συμφωνιών από την πλευρά της νέας Αμερικανικής κυβερνήσεως και πώς θα συνεργαστούμε. Νίνα Γκίλ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Χαίρομαι για τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν σχετικά με τον ΝΑΤΟ στην συζήτηση. Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηγέτης στην χορήγηση ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας. Δεν θα πρέπει να λησμονείται αυτό. Όταν δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείε εξαρτούν τη συμμετοχή του στο ΝΑΤΟ από την αύξηση των συνεισφορών των ευρωπαϊκών χωρών μέλων. Α μην λοιπόν αυτό. Ένα χώρο στον οποίο αναφερθήκατε ήταν η Ασία. Και σε σχέση με το πού μπορούμε να συνεργαστούμε. Πρόκειται για μια περιοχή του κόσμου που αντιμετωπίζει σοβαρότατες απειλές στην ασφάλεια και ιδίω στην θάλασσα, αλλά βεβαίως και από την Βόρεια Κορέα. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν περισσότερα για την Ασία και πού βλέπετε, σε ό,τι αφορά την Βόρεια Κορέα, πού βρίσκονται οι απαράβατες ερυθρές γραμμές το ίδιο για την ασφάλεια στη θάλασσα, νότια κινέζικη θάλασσα, που βρίσκεται εκεί πάλι ε, η απαράβατη γραμμή σας. Θεωρείτε ότι υπάρχει χώρος συντονισμού Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένης Ευρώπης και θεωρείτε ότι μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι σημαντικοί ε, παίκτες από την Ασία, για παράδειγμα οι Ινδίες. Η κυρία Φώτιγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Πρέσβη στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Μου φάνηκε πολύ ξεκάθαρη και καθησυχαστική η δήλωσή σας. Δεν έχω λοιπόν μείζωνα σχόλια, πάντως εκφράζω την εκτίμησή μου για την προωθημένη παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στο, στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης, πολύ σημαντικό για εμάς τους Πολωνούς. Η Πολωνία επιθυμεί να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή. Και θα συμμετέχουμε στις επιχειρήσεις και στην Λετωνία και αλλού. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε λίγα περισσότερα για τις εξελίξεις για τον ε, παγκόσμιο συνασπισμό κατά του ISIS. Και δεύτερο, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος προσεγγίσεως για την ολοκλήρωση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά ασφάλεια και άμυνα. για να εξασφαλιστεί έτσι η ορθή συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Αργίζει και παίρνει χαρακτήρα πραγματική ακρόαση η συνεδρίαση, λέει ο πρόεδρο Μακάριστερ. Από την Ενωτική Αριστερά, ο κύριος Κόουσο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι πολύ καλό που μπορούμε να έχουμε μια πρώτη επαφή με τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ. Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Η απειλή η ρωσική είναι της μόδας έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μην ανησυχείτε. Για τον ΝΑΤΟ λοιπόν. Για την δικιά μας ε, ικανότητα στην Ευρώπη και οι δαπάνες στην άμυνα μας ε, ζητούν να δαπανούμε περισσότερα παρά την ε, σοβαρή κρίση μέσα στην οποία βρισκόμαστε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αν μη τι άλλο στην περιφέρεια της Ευρώπης που υποφέρουν από τη λιτότητα. Αυτά που είπατε για το Ιράν με εκπλήσουν, γιατί είπατε ότι από εκεί απορρέει σε ένα μεγάλο βαθμό η τρομοκρατία. Ε, Συρία, κάποιοι σύμμαχοι της χώρας σας και της δικιάς μου δυστυχώς και αυτοί φέρνουν όμως τρομοκρατία. Οπότε ρωτάω, με το Γουαντάναμο τι θα κάνει η κυβέρνησή σας. Υπήρχε μια υπόσχεση ότι θα κλείσει επειδή ήταν εκτός του κράτους ε, δικαίου. Θα το τηρήσει ο πρόεδρος και η Σύρια. Θα υπάρξει συμφωνία με την Ρωσία για να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα εκεί. Και για τον ΝΑΤΟ θα σταματήσετε να συνεισφέρετε όπως το κάνατε μέχρι τώρα. Τι σχέση θα έχετε με τον ΝΑΤΟ, θα συνεχίσετε να συμμετέχετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε ή θα απαντήσετε. Ας ακούσουμε και την κυρία Λούνατσεκ εκ μέρους των Πρασίνων για να έχουμε κάνει τον γύρο των ομάδων. Ευχαριστώ και εκ μέρους των Πρασίνων σας ευχαριστώ που ήρθατε για να έχουμε τη συζήτηση αυτή μαζί. Λοιπόν, κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε μέχρι τώρα. Ναι, μιλάτε πολύ για την ασφάλεια για τους Αμερικανούς πολίτες. Λέτε επίσης ότι θέλετε να συνεχίσετε να στηρίζετε τον ΝΑΤΟ, τη συνεργασία μας κτλ. Αλλά όταν αναφέρεστε στην ασφάλεια σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Υπάρχει κλιματική αλλαγή, Υπάρχει το θέμα του πώς θα συνεργαστούμε με αναπτυσσόμενες χώρες. Και από αυτά που ακούσαμε πρόσφατα θα υπάρξουν περικοπές. Ένα τρίτο στα κονδύλια ε, του Υπουργείου Εξωτερικών για προγράμματα, για συνεργασία ε, με χώρες που προσπαθούν ε, να αμβλύνουν την κλιματική αλλαγή. Είδαμε πλημμύρες σε ένα σωρό σημεία του κόσμου που έχουν να κάνουν με την ε, ανθρωπογενή δράση που οδηγεί στην κλιματική αλλαγή. Επίσης, είπατε ότι θα μειωθούν τα κονδύλια και για τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα. Και αυτό είναι όμως κάτι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών. Οι περικοπές των 600 εκατομμυρίων που θα κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείες πρόκειται για 6,5 εκατομμύρια παραπάνω ε, εγκυμοσύνες που δεν θα παρακολουθούνται, για παράδειγμα, ή όσες αμβλώσεις. Οπότε θέλω να ξέρω, υπάρχει περίπτωση οι περικοπές αυτές στην εξωτερική συνεργασία και για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι να μην υλοποιηθούν ως περικοπές. Ωραία. Ολοκληρώνεται με τον κύριο Καστάλτο ο πρώτος γύρος παρεμβάσεων. Παρακαλώ κύριε Καστάλτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Σουμπ για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις τους. Στις ερωτήσεις μου θα, θα αναφερθώ στις νέες στρατηγικές προτεραιότητες του Λευκού Οίκου όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Είπατε ότι το Ιράν είναι βασικός υποστηρικτής των τρομοκρατών. Εγώ μπερδεύομαι διότι σχεδόν οι τρομοκρατικές όλες οι ομάδες είναι σουνητικές. Άρα μου φαίνεται λίγο περίεργος ορισμό αυτός. Πέραν από αυτό θα ήθελα να ξέρω να περιμένουμε λοιπόν ότι θα συζητηθεί συμφωνία για τα πυρηνικά. Αυτή η συμφωνία τελικά θα αμφισβητηθεί από τη νέα κυβέρνηση στη Συρία. Ποια είναι η προτεραιότητα στρατηγική όσον αφορά την κατάληψη της ΡΑΚΑ. Πώς βλέπετε τη συνεργασία τη Αμερικανική κυβερνήσεω με άλλου φορεί περιφερειακού και παγκόσμιου που είναι παρόντε στη σκακέρα τη Συρία. Και άλλη μια ερώτηση που αφορά το ρόλο τη Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή γίνεται πάρα πολύ αυταρχική εν αναμονή αυτού του συνταγματικού δημοψηφίσματο. Ποια είναι η θέση σα όσον αφορά το ρόλο που παίζει εντό του ΝΑΤΟ η Τουρκία. Μια άλλη ερώτηση που αφορά την Κούβα. Επανειλημμένα είδαμε τον πρόεδρο τον κύριο Τραμπ κατά κάποιο τρόπο να αποστασιοποιείται από τα ανοίγματα που έγιναν την προηγούμενη κυβέρνηση του κύριου Ομπάμα. Θέλουμε να καταλάβουμε λοιπόν ποιε θα είναι οι θέσει τη κυβερνήσεω τη Αμερικανικής όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Κούβα και ΙΠΑ. Τι να περιμένουμε εκεί. Τέλος, μια άλλη ερώτηση κλείνοντας. Όσον αφορά την Κίνα. Πριν αναφερθήκατε στη στάση της ε, συστάσει της έναντι της και το κόστος της παγκοσμιοποίησης, κάτι που μας ευαισθητοποιεί. Ποια θα είναι η στάση σας. Θα υπάρξει κάποια εντό εγωγικών αντιπαράθεση εμπορική με το Πεκίνο ή θα τηρηθούν υποσχέσεις μιας, ενός αγώνα δρόμου εξοπλισμών όπως είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση προεκλογικά ε, όσον αφορά την απέναντι στην Κίνα. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ο Πρόεδρος. Άντα, πολλές και διάφορες ερωτήσεις. Μέχρι το βράδυ θα μπορούσαμε να μείνουμε εδώ. <clears throat> Απαντήστε στον πρώτο γύρο και να ξέρουμε ότι έχουμε άλλους 11 συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο κλείνει ο κατάλογος ομιλητών. Έτσι δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους στον κατάλογο. <clears throat> Τόσες πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, σας ακούμε για την απάντησή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν ε, δεν σας πειράζει, θα συγκεντρώσω ένα θέμα. Τις ερωτήσεις για να απαντήσω ένα θέμα. Για κάποια πράγματα δεν έχουμε απαντήσεις. Για το μου για την Κούβα μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μια αναθεώρηση που πραγματοποιείται, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Οπότε δεν είμαι σε θέση να σας πω ποια θα είναι η πολιτική μας. Ας έρθω στην Κίνα. Στο εμπορικό πλαίσιο μιλούμε για την Κίνα. Είμαστε στο ίδιο σημείο νομίζω και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε καλωσορίζουμε τα εμπορικά ανοίγματα της Κίνας, συμμετοχή στο G20, αλλά πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί για πράγματα όπως είναι οι επενδύσεις. Το είδατε και οι ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να εξετάζουν πιο στενά τις κινέζικες επενδύσεις. Τώρα, ο Υπουργό Εξωτερικών ήρθε από την Απανατολή πρόσφατα. Η κυβέρνησή μας σκοπεύει να συνεχίσει επικοδομητικές σχέσεις με την Κίνα. Συγχρόνως όμως θα διασφαλίσει, θέλει να διασφαλίσουμε ότι η Κίνα θα τηρεί τους διεθνείς κανόνες για το εμπόριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Ο πρόεδρος ε, Τραμπ έχει μιλήσει με τον ε, κύριο Σι και νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούν στη Φλόριντα. Συμφώνησαν ε, λοιπόν οι δύο ότι υπάρχει περιθώριο για περισσότερη συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών και αποφάσισαν να ενισχύσουν τις σχέσεις. Οπότε υπάρχει περιθώριο για συνεργασία, προσπάθειες θα συνεχιστούν, αλλά παρακολουθούμε συγχρόνως το οικονομικό σκέλος, το εμπορικό και τον ρόλο που παίζει η Κίνα στην νότια Κινέζικη θάλασσα και τη σχέση της με τις γειτονικέ της χώρες, Φιλιππίνες, Βιετνάμ, είναι πράγματα που μας απασχολούν σοβαρά. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ λίγο και στη Βόρεια Κορέα. Υπάρχουν σε βάθος συζητήσεις που έγιναν από τον Υπουργό μας με την κινέζικη κυβέρνηση προσπαθούν να δούνε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα για αυτά, δεν έχω περισσότερα. Έρχομαι τώρα στο εμπορικό σκέλος, εμπόριο. Η πέτροπος Μάλστρομ αναφέρθηκε στο TTIP λέγοντας ότι έχει μπει στο ψυγείο. Νόμιζα κι εγώ ότι είχαμε δυόμιση χρόνια επικοδομητικών διαπραγματεύσεων στις οποίες ε, συζητήθηκαν ερωτήσεις όπως αυτές που θέσατε εδώ σήμερα το TTIP θα μπορούσε, έτσι το είχαμε δει και οι δύο πλευρές, να είναι μια συμφωνία υψηλών προδιαγραφών. Έχει να κάνει με τους δασμούς, με τις υπηρεσίες, με τις συνθήκες εργασίας, με ένα σωρό πράγματα. Η σχέση αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές στον κόσμο. 4,5-3 δολάρια επενδυτική σχέση 25 δις όσον αφορά τις αμερικανικές εξαγωγές από μόνες τους. Πρόκειται επίση για συναλλαγέ μεταξύ των εταιριών κατά το ανατρίτο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τι εταιρείε μα εκατέρωθεν. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Ξέρετε ποια είναι η θέση του Πρόεδρου για το TTIP. Αλλά το TTIP δεν είναι σε μια ειδική κατηγορία. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε ακρόαση του εμπορικού επιτετραμένου, πήγε καλά και όταν θα οριστεί ε, τελειωτικά θα ξέρουμε περισσότερα. Υπάρχουν θέματα και στον ε, ΠΟΕ που προχωρούν θετικά. Πριν από τρεις εβδομάδες υπογράψαμε συμφωνία για το MRA, έτσι το λέμε νομίζω. Είναι συμφωνία για πρακτικές μεταποίησεις στην φαρμακοβιομηχανία. Γίνονται τώρα συζητήσεις ανά τομέα, οπτικοακουστικά, στο εμπόριο. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε οικονομίες από τις επιχειρήσεις και στον ΠΟΕ, ναι, υπάρχουν υποθέσεις του ενός εναντίον του άλλου, αλλά προσπαθούμε να καθορίσουμε ένα σύστημα κανόνων που να αφορά όλους, και τους νέους και τους παλιούς. Οι πολυμερείς συμφωνίες μας ενδιαφέρουν όλους ιδιαίτερος. Το Buenos Aires ξέρετε ότι θα έχει σύντομα μια υπουργική συνάντηση για το εμπόριο. Για τον προπολογισμό δεν έχω πολλές απαντήσεις. Όπως ξέρετε, καλύτερα εσείς από οποιοδήποτε άλλον, ο προπολογισμό χρειάζεται μακρές διαπραγματεύσεις. Και το μόνο που έχουμε δει από την κυβέρνηση προς το παρόν είναι έναν αδύναμο προπολογισμό. Είναι δύσκολο να πούμε πού πάμε. Συνάδελφοί σας και άνθρωποι με τους οποίους έχετε συναντηθεί έχουν σχολιάσει για το πώς θα ψηφίσουν για τον προπολογισμό. Ε, αυτή δεν είναι δικιά μου δουλειά εδώ να σχολιάσω ή να κάνω υποθέσεις για το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση με τον προπολογισμό, σίγουρα είναι δύσκολο να καταλήξουμε στον προπολογισμό. Και δεν είναι κάτι νέο, δεν οφείλεται στη νέα κυβέρνηση Τραμπ και άλλες κυβερνήσεις δυσκολεύτηκαν να καταλήξουν στον προπολογισμό τους. Και δεν ξέρω ποιος το έχει πει, αλλά νομίζω ότι μετά από κάθε συζήτηση που γίνεται για τον προπολογισμό στο Καπιτόλιο, ε, λέμε ότι χύθηκε αίμα τελικά και τα μέλη του Κογκρέσου και οι γερουσιαστές έχουν πράγματι έντονες συζητήσει. Για το θέμα της Τουρκίας. Νομίζω ότι ανησυχούμε και εσείς και εμείς για τέτοια πράγματα. Αλλά να πω πρώτα απ' όλα ότι είναι μια δυνατή χώρα σύμμαχος η Τουρκία, κοντά στην ε, ε Μέση Ανατολή, ισχυρός σύμμαχος που έχει αναλάβει το βάρος της μετανάστευσης γιατί είναι ανάμεσα στην Συρία και τους υπόλοιπους, όλα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Αλλά και εμείς εκφράζουμε ανησυχίες. Και έχουμε πει στους Τούρκους και δημόσια αλλά και ιδιαίτερος ότι το θέμα των ελευθεριών των πολιτών, των πολιτικών δικαιωμάτων, της ελευθερίας ε, τύπου, ακόμα και οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί. Είπαμε λοιπόν ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Αντιλαμβανόμαστε ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, κρίσιμο στην επίλυση της μεταναστευτικής κρίσης. Τους ενθαρρύνουμε να είναι επικοδομητικοί και να είναι επικοδομητικοί και στο θέμα της Κύπρου. Βασίζουμε πολλές, μάλλον βασίσαμε πολλές ελπίδες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Τουρκία μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και συνομιλίες έχουμε, όπως σας είπα, και, σε, και δημόσιες αλλά και σε ιδιωτικό επίπεδο μαζί τους. Συρία. Συρία. πραγική κατάσταση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είμαστε στον 7ο χρόνο της κρίσης αυτής και ο κόσμος υποφέρει όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Δεν έχουν τρόφιμα, νερό, βασανίζονται, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ο μισός πληθυσμός έχει φύγει από τα σπίτια του, τα παιδιά, είναι μεγάλη τραγωδία. Εμείς κάθε φορά που μπορούμε επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για ειρήνευση. Στηρίζουμε τον ΟΙΕ, τον εκπροσωπό, το έχουμε και το δικό μας, τον Μακλιράντνε εκεί, για να διευκολύνουμε το διάλογο, να υπάρξει πολιτική λύση βάσει της οποίας να ανακτηθεί η ειρήνη και η σταθερότητα για τον κόσμο εκεί και να μην υπάρχει πια απειλή της τρομοκρατίας. Προς το σκοπό αυτό λοιπόν μπορώ να πω ότι με ικανοποίηση θα συμμετάσχουμε σε τρεις εβδομάδες στη διάσκεψη για την ειρήνευση στη Σύρια. Εδώ στις Βρυξέλλες θα είναι μια καλή ευκαιρία, το κουαρτέτο δηλαδή συμμετέχει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και οι ανθρωπιστικές ανάγκες Στη Γενέβη βέβαια πρέπει να υπάρξουν συνομιλίε. Αυτό είναι ο κατάλληλο τρόπο, αλλά βέβαια δεν μπορεί κανεί να αντιμετωπίζει το θέμα ή όλα ή τίποτα. Ήμασταν και στην Αστάνα ω παρατηρητέ πριν από λίγο καιρό. Πιστεύουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, ήταν εκεί και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε για να λυθεί αυτό το θέμα. Τώρα το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής Υπάρχουν ε, διάφορα προγράμματα υπέρ των γυναικών, επειδή είπατε ότι θα τα σταματήσουμε. Είναι πολύ σημαντικά. Είναι σημαντικοί παράγοντες όλα αυτά όταν εξετάζουμε το θέμα της σταθερότητας, σταθερότητας των κοινωνιών και την ευημερία του κόσμου, εννοείται ότι τα εξετάζουμε αυτά βέβαια. εξαρτάται πώς ε, και από ποια πλευρά κοιτάζει κανείς τα πράγματα. Σίγουρα υπάρχει πολλοί κόσμος σε φτώχεια, σε προσφυγιά και τα λοιπά που πρέπει να βοηθηθούν. Αλλά υπάρχουν πολλές απειλές. Υπάρχουν στρατιωτικές απειλές που μας έρχονται εξ Ανατολών, που πρέπει να αντιμεταπιστούν και πολλές από τις δικές σας χώρες συμμετέχουν στον συνασπισμό και στρατιωτικά. Οι στρατιωτικές απειλές λοιπόν επίσης πρέπει να αντιμετωπιστούν στρατιωτικά. Μετά θα δούμε το θέμα της αποκατάστασης, της ανοικοδόμησης. Το ξέρει η κυρία Μογκερίνη, το συζητάμε και μαζί της και ελπίζω να πετύχει διάσκεψη για τη Συρία που θα γίνει εδώ σύντομα. Νομίζω ότι αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ για αυτό τον πρώτο γύρο. Συνάδελφοι, προτείνω να μειώσουμε το χρόνο αγόρευσης 1,5 λεπτό. ρωτήστε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν. Κύριο Σαλαφράνκα για το ΕΛΚ είναι επόμενος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Κύριε Πετετραμένα. Θαυμάζω πολύ τις Ηνωμένε Πολιτείες που μπορεί και παράγει το 25% αγαθών και υπηρεσιών όμως τα μηνύματα από την κυβέρνησή σας δεν είναι πολύ φιλικά. Η πρώτη επένδυση είπατε ότι η κυρία Μάρστρομ είπε ότι το τύπη πήκε στο ψυγείο. Ε, εσείς ε, είπατε πράγματα θετικά μερικές φορές για το Brexit, επικρίνατε διάφορες χώρες. Η καγκελάριος και οι Πρωθυπουργό πήγανε στι Ηνωμένε Πολιτείε ήδη και συναντήθηκαν με την Αμερικανική κυβέρνηση. Να ξέρετε ότι πολλές από τις δηλώσεις που ακούγονται ανησυχούν τους πολίτες. Συνεπώς, θα ήθελα να διαλύσετε κάπως τις αμφιβολίες που υπάρχουν όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τη στάση της κυβέρνησή σας. Όπως επίσης όσον αφορά την πολυμερή διάσταση, ε, επειδή αναφέρθηκε ο πρόεδρος στο, στη σχέση με τον ειρηνικό πιο πολύ. Και θέλω και κάτι άλλο που είναι πολύ της μόδας στη σχέση μας με τις ΗΠΑ, που είναι η Ρωσία. Στην Ολομέλεια, όταν είχαμε τη συζήτηση για το Μαυροβούνιο, συζητήσαμε και γι' αυτό. Υπάρχει κάποια δραστηριότητα επ' αυτού. Και τέλος, η θέση σας για την Άπο θα συνεχίσει στην ίδια Ευχαριστώ κύριο Πάσκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πολυμερές δίκτυο εμπορικών συμφωνιών συμμετέχει στην ε, ειρήνευση και σταθερότητα στον κόσμο. Αυτό αγνοείται ή υποτιμάται, αλλά είναι θεμελιώδου σημασία σε αυτές τις συμφωνίες για την ειρήνη και σταθερότητα του συστήματος. Και για τα 70 χρόνια μετά το αυτό το πόλεμο η συνεισφορά αυτών των συμφωνιών ήταν ε, τεράστια. Όλοι ξέρουμε ποιε είναι οι σκέψει τη νέα κυβερνήσεω για σημαντικά τμήματα του δικτύου αυτού. Αλλά ερώτηση. Κατά την άποψή σα, αυτό αντικατοπτρίζει νέα φιλοσοφία τη κυβέρνηση και αφορά όλο το δίκτυο των συμφωνιών είναι κάτι που αφορά ξεχωριστές συμφωνίες, διότι το σωρευτικό αποτέλεσμα των διαφόρων κομματιών υπονομεύει το δίκτυο. Το γνωρίζει αυτό η κυβέρνηση ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ κύριε Πάσκου. Τσάρλς Τάνοκ για το ECR. Ευχαριστώ. Διαδικαστικό. Δεν μου δόθηκε ο λόγος να μιλήσω σαν συντονιστής του ECR όταν δόθηκε ο λόγος σε κοσόπου της ομάδας. Θα είμαι σύντομος. Ευπρόσδεκτα τα θετικά μηνύματα από τη Ουάσιγκτον. Άρα τα διάφορα λόγια της προεκλικής η ενθάρρυνση του Brexit, η κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η υπονόμευση του ΝΑΤΟ, όλα αυτά μάλλον αποτελούν παρελθόν όπως υπόθηκε και στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου και στις Βρυξέλλες, αυτά υπόθηκαν καθιστικιστικά. Κρυγονίως λήθος για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι ε, η ΕΠΑ και για το εμπόριο και την ασφάλεια και για τις σχέσεις με την Βρετανία μετά τον Brexit. Λυπηρό, ο θάνατος του TTIP και η απόσυρση από τη Συμφωνία του Ειρηνικού και η από τη Συμφωνία των Παρισίων. Λυπηρό διότι θα υπάρχουν ε, μαζικές μεταστευτικές ροές στο μέλλον αν δεν συγκρατήσουμε τις, τα αποτελέσματα της αλλαγής του κλίματος, κυρίως όσον αφορά την υποσαχάρια Αφρική. Υποστηρίζω την άποψή σας. Το Ιράν θα πρέπει να εμποδιστεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Θα πρέπει να μας στηρίσει την τήρηση της συμφωνίας και θα πρέπει να συνεχιστούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την, το θέμα της Κρυμαίας και θα πρέπει να συμμορφωθεί η ψηφορία του Μίνσκ. Για το Κυρκούκ θα υποστηρίξετε τους Κούρδους. Ευπρόζεκτο αυτό. Και θα είσαστε και φιλικοί έναντι της δημοκρατίας της Κίνας. Και τελικά πρέπει να ιτηθεί και το ISIS και να σταθεροποιηθεί η Συρία. Λατινική Αμερική τι γίνεται. Με το Μεξικό τι θα γίνει με το τείχος με το Μεξικό. Που είναι επίμαχο θέμα. Και θέλουμε να δούμε θα είναι Τέντ Μάλοχ ή άλλο. Θέλουμε να δούμε ποιος θα είναι ο νέος πρεσβευτής ε, των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Χατζηγεωργίου είναι επόμενο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συντομότατα ερωτήσεις, ε, ερωτήματα. Δύο τον αριθμό. Που απευθύνω στον εκπρόσωπο τον είπα, τον κύριο Πρεσβευτή. Πρώτη ερώτηση. Ο κ. Ερντογάν ζήτησε η χώρα του να είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σαν Ισλαμική χώρα, είπε. Σαν μουσουλμανική χώρα. Έχετε κάποια αντίδραση γι' αυτό. Ποια είναι η απόψη σας. Δεύτερον, αναφερθήκατε στο Κυπριακό. Ξέρω ότι γνωρίζω ότι δεν εξάγονται συζητήσεις τώρα. Οι διαπραγματεύσεις έχουν διακοπεί. Έχετε κάποια γνώση ε, γιατί συνέβη αυτό. Έχετε παίξει κάποιο ρόλο πάνω σε αυτό. Θα παίξετε κάποιο ρόλο πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ κύριο Κάβα για το EFDT. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χάρηκα για τα σχόλιά σας. Είπατε ότι πρέπει να είναι πυλών σαμινάς μας στο ΝΑΤΟ. Καλό αυτό. Ε, οι στατιωτικέ φιλοδοξίε τη Ευρωπαϊκή Ενώση πώ επηρεάζουν τον ΝΑΤΟ και τι μελλοντικέ δεσμεύσει των ΗΠΑ. Όσον με τον Brexit. Θα υπάρξει πιο στενή στατιωτική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου εκτό των διεθνών θεσμών. Δεν αναφερθήκαμε στο Ισραήλ. Τέτοια απόκληση απόψεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και ΗΠΑ υπάρχει όσον αφορά το Ισραήλ. Υπάρχουν διαφορέ, άρα μπορεί να υπάρχει κοινή προσέγγιση όσον αφορά το Ισραήλ. Μετά η Εμένη. Καταστροφική κατάσταση στην Εμένη. Επικρατεί αστάθεια. Σε μια ευμετάβλητη περιοχή. Η ΙΠΑ θα παίξουν αυξανόμενο ρόλο στην περιοχή. Κυρίω να αφορά τι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνεχίζονται. Τέλο. Πρόεδρο Τραμπ. Η Ουάσιγκτον πώ βλέπει τα σχόλια τα υποτιμητικά που ακούγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του κυρίου Τραμπ και κάποιοι ε, βουλευτές Ευρωπαίοι. Ε, όπως και να τον εμποδίσουν να, να εκφράζει την άποψή του, να μιλήσει, να κάνει ομιλίες. Η κυρία Μανέσκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Σούμπ στη συνάντησή μας. Πολύ σημαντική ανταλλαγή απόψεων. Πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να τεθεί τέρμα στην προεκλογική ρητορική. Δεν είναι επικοδομητική ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε για τη ΣΥΠΑ, ούτε για τις σχέσεις μας. Βοηθά μόνο τους ε, μη φίλους μας, όπως η Ρωσία. Οι σχέσεις μεταξύ μας είναι πολυσχηδείς. Χρειάζεται ρεαλιστική προσέγγιση. Να εξετάζουμε κάθε πτυχή. Διεθνείς σχέσεις όσον αφορά την ασφάλεια και το ΝΑΤΟ είναι σημαντικά αυτά τα θέματα. Κάθε χώρα πρέπει να πληρώνει το λογαριασμό της. Η Ρουμανία, η πατρίδα μου, είναι μία από τις πέντε χώρες που πληρώνει αυτά που πρέπει. Περιμένουμε και άλλοι να κάνουν αυτά που πρέπει. Η Ρωσία και η συμπεριφορά της όσον αφορά την Ουκρανία. Άλλο κοινό μας πρόβλημα προς επεξεργασία. Έχω μεγάλες προσδοκίες όσον αφορά τα αποτελέσματα μετά το διορισμό της κυρίας Φιώνα Χιλ, που θα είναι ένα από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ερώτηση. Τι να περιμένουμε από την κυβέρνηση, από πλευράς αποφάσεων και δράσεων, για τη σχέση με το Ιράν, εξομάλυνση σχέσεων με τη Ρωσία και καταπολέμηση τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ραμόνα. Ο κ. Φρόιντ για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σουμπ που παρίσταστε. Χαίρομαι για αυτά που είπατε. Χαίρομαι επίσης ότι μας καθησυχάσατε. Μιλήσατε σαν να μην άλλαξε η κυβέρνηση στη Ουάσιγκτον, σαν να μην άλλαξε κάτι. Ε, είδα τις αλλαγές από τον Τζίμι Κάρτερ μέχρι τον Ρέιγκαν. Όμως, ποτέ δεν είδα αλλαγή σαν την τωρινή. Και αυτά που είπε και ο κύριος Τρόμπ για τον προκάτοχό του δεν θέλω καν να τα επαναλάβω. Σκέφτομαι τι θα λέει και για από τους συμμάχους του στην Ευρώπη ο κύριος Τραμπ. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι ο Νάιτζελ Φαράζ ήταν ένας από τους πρώτους που του ψιθύρισε στο αυτή τι, περιτίνος, για το τι περιτίνος πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ποιος άλλος τον συμβουλεύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αντιμετωπίζει τη ΣΥΠΑ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από την Άγγελα Μέρκελ που πήγε προημερών βέβαια. Αυτή είναι μία ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Οι νέοι κανόνες για, τα, για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό για κάποιες μεσανατολικές χώρες. Ισχύει κάτι τέτοιο για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, αυτό που ισχύει για τις μεσανατολικές χώρες. Ο κύριος Γιούρεκ για το ECR. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, φορέστε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις. Ευαίσθητα θέματα αφορούν για την περιοχή μας. Κυρίως για τους συμμάχους μας που είναι πιο ευάλωτοι και απειλούνται. Εστονία, Λετωνία. Οι ΙΠΑ θεωρούν ότι εξής τον κόπο να ενισχυθεί η ασφάλειά τους περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το τι συνέβη τον τελευταίο χρόνο. Δεύτερο ερώτημα, Γεωργία. Σε σχέση με την Κρυμαία, η Γεωργία είναι άλλη μια χώρα που θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα κάποιο σχόλιο για τις ελπίδες και τις απειλές για αυτές τις χώρες. Πρέπει να ενισχυθεί η ασφάλεια της Γεωργίας, πιστεύω. Πρέπει να γίνει σύμμαχός μας ή τουλάχιστον να πούμε ότι υπάρχει κάποια πρόθεση τέτοια. Θέλω να εκφράσω επίσης την έγκρισή μου για την απόφαση του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το να σταματήσει η χρηματοδότηση για τις αμβλώσεις στον κόσμο. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις γι' αυτό στο Κοινοβούλιο. Εκατομμύρια όμως Ευρωπαίοι θεωρούνται ότι ε, υποεκπροσωπούνται και θεωρούν ότι αυτή είναι πραγματική κίνηση για αποκατάσταση της ηθικής τάξης και της ηγεσία σε ηθικά θέματα, τον είπα, στον κόσμο. Σύμφωνα με την παράδοση, οι Αμερικανοί πρέπει να γνωρίζουν ότι και στην Ευρώπη έχουμε παρόμοιες απόψεις. Ευχαριστώ. Οι τελευταίοι τρεις. Πρώτος ο κύριος Γκάλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. η πρώτη μου ευχή προς εσάς κύριε Επιτετραμένε είναι να υποδεχθείτε τον νέο πρέσβη και να είναι το ίδιο καλός όπως ο προηγούμενος Αμερικανός πρέσβης εδώ. Έχοντας τώρα υπόψη την ε, διάσκεψη ασφάλειας του μονάχου. Με καθησύχασαν ο αντιπρόεδρός σας και ο Υπουργός Άμυνας και ιδίω με εντυπωσίασε η δικοματική ομάδα του Κογκρέσου και ο τρόπος με τον οποίο συμμετέσχουν στις συζητήσεις και έχοντας ακούσει τις προθέσεις τους σχετικά με τη Ρωσία και τι σχεδιάζουν για φέτος, η ερώτηση που αναπηδά είναι η εξής. Μπορεί να υποθέσει κανείς ότι η πολιτική απέναντι στη Ρωσία προωθείται περισσότερο από το Κογκρέσο και λιγότερο από το State Department και ακόμα λιγότερο από το Λευκό Οίκο, όπου ακόμη δεν είναι σαφές ποιοι ακόμη έχουν από τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου κάποιες σχέσεις με τη Ρωσία. Η άλλη πτυχή, σε ό,τι αφορά ασφάλεια και άμυνα, καθώς ξεκινούμε να αναλάβουμε ακόμα περισσότερα εδώ στην ευρωπαϊκή πλευρά, μπορεί, νομίζετε, να αντιληφθεί η νέα Αμερικανική κυβέρνηση ε, περισσότερο τα πράγματα αυτά όπως συνεργασία, κοινό σχεδιασμό, κοινέ προμήθειε, που όλα αυτά επίση ενισχύουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Και ποια είναι η πιθανή απάντηση της νέας Αμερικανικής κυβέρνησης. Ελπίζω μάλιστα να είναι η ίδια όπως αυτή που είχε δοθεί από την προηγούμενη Αμερικανική κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Τώρα εσείς κύριε Μποστινάρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτετραμένε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που συμμετέχω στη συζήτηση. Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Πρώτη, ποιος είναι ο ρόλος και πόσο περιθώριο συνεργασίας και συντονισμού υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ηνωμένων Πολιτειών για τη Ρωσία και ιδιαίτερα για τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Επειδή είναι γνωστό ότι το θέμα αυτό θα επανέρχεται ανά Δεύτερο, Γνωρίζετε ότι μετά από την Συρία η Ρωσία έχει αναπτύξει δύο μέτωπα. Ένα στην Ανατολική Μεσόγειο και ένα προς την Μαύρη Θάλασσα. Επιτρέποντας την πρόσβαση και απαγορεύοντας την πρόσβαση. Που σημαίνει ότι είναι αναγκαία μια ιδιαίτερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ γενικότερα. Πώς το βλέπετε αυτό. Και τέλος, ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των ΗΠΑ στον ειρηνικό, γνωρίζοντας ότι η απόφαση να αποσυρθούν από τη συμφωνία TPP δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η κινέζικη κυριαρχία στον ειρηνικό. Ευχαριστώ. Τούνε Κέλαμ. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής. Χαίρομαι για την παρουσία σας εδώ ενώπιόν μας. Να πω ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή στην πιο στενή ε, διατρατική συνεργασία. Είμαι εστονός και θεωρώ ότι μας καθησυχάζουν πολύ, και το λέγω, η παρουσία των Αμερικανικών δυνάμεων στα ε, ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Ταυτόχρονα η εξοπιστία του ΝΑΤΟ αμφισβητείται στην περιοχή αυτή του κόσμου. Ερώτηση, είστε διατεθειμένοι και να αντιμετωπίσετε υβριδικές μορφές εισβολής, διότι αυτό αποτελεί μέρος των ρωσικών δραστηριοτήτων. Δεύτερο, χρειαζόμαστε στενότερη συνεργασία για υποστήριξη της Ουκρανίας απέναντι στις δραστηριότητες των Ρώσων. και ενδεχομένως και χορήγηση αμυντικών όπλων στην Ουκρανία. Τρίτο, Ποια είναι η εκτίμησή σας σχετικά με τον ρόλο του Ιράν ως παράγοντα αποσταθεροποίησης, διότι το Ιράν είναι μέρος του προβλήματος βεβαίως και όχι της λύσης. Και οι δύο πλευρές ωστόσο έχουμε προκαλέσει το κενό στην Μέση Ανατολή, το οποίο κενό πληρώθηκε από Ρωσία και Ιράν. Είπατε ότι οι στρατιωτικές απειλές πρέπει να αντιμετωπίζονται με στρατιωτικά μέσα. Μπορεί ωστόσο εδώ να υπάρξει κάποια κοινή προσέγγιση στα προβλήματα που σημειώνονται στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Μακάριστερ, ευχαριστώ πολύ για τις ε, ερωτήσεις σας που και πάλι καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων. Θα σας δώσω 15 λεπτά για να απαντήσετε σε όσο μπορείτε περισσότερες από αυτές. Ευχαριστώ αγαπητέ πρόεδρε. Να απαντήσω σύντομα. Για την Κύπρο. Είμαστε φίλοι και της Ελλάδος και της Τουρκίας. Και αυτός είναι ο ρόλος μας. Είμαστε σύμμαχοι και των δύο αυτών χωρών. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι οι συνομιλίε δεν προχωρούν. Έχουμε ένα αριθμό αξιωματούχων που έχουν έρθει εδώ, έχουν πάει και στην Άγκυρα, έχουν πάει και στη Λευκοσία και βεβαίω και, και στην Αθήνα για τι σχετικέ συζητήσει. Βρισκόμαστε λοιπόν συζητήσει για το μέλλον τη Κύπρου, που βεβαίω και αυτό είναι ένα, ένα πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο θέμα και το οποίο συνεχίζεται. Να μιλήσω λίγο περισσότερο για τη Ρωσία, διότι είναι κρίσιμο θέμα για όλου μα. Μια Ρωσία με επιθετικές δράσεις και στην Ανατολική Ευρώπη και απέναντι στι Ηνωμένες Πολιτείε, αλλά και παραπέρα από αυτά όπως είδαμε στις σημερινές ειδήσει και που δεν δείχνει σημάδια αλλαγής πορείας. Τα είδαμε και στη Συρία, είδαμε όπως είπα και στις ειδήσει σήμερα το πρωί, αναφέρομαι δηλαδή στις στρατιωτικές δραστηριότητες. Αυτό τονίζουν άλλωστε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι και στις συζητήσεις τους με Ευρωπαίους συμμάχους, αλλά και ο Υπουργό Εξωτερικών Τίλερσον θα συναντηθεί τότε την εβδομάδα πιθανότατα με όλους τους υπουργούς, Εξωτερικών στην ε, στην Ουάσιγκτον πολλούς από τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και μια μεγαλύτερη ομάδα υπουργών εξωτερικών. Είναι απολύτως ε, αναγκαίο, είναι επιτακτικό και αυτή ήταν και η πολιτική της προηγούμενης Αμερικανικής κυβερνήσεως και αυτά ακούσαμε και από τον Υπουργό μας των Εξωτερικών, αλλά και τον Υπουργό Άμυνας και από τον Σύμβουλο Εθνική Ασφαλεία. Είναι αναγκαίο οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργάζονται απέναντι στη Ρωσία, απέναντι σε τόσα πολλά θέματα. Στρατιωτικά, βλέπει Ουκρανία, ε, Μέση Ανατολή, και βεβαίως και πώς να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά αυτό τον μη γραμμικό πόλεμο, υβριδικό ε, πόλεμο παραπληροφόρησης, επιρροή εκλογών που ε, θίγει και την Ευρώπη, θίγει και τις Ηνωμένες Πολιτείες όπως γνωρίζετε. Έχουμε λοιπόν κάποια ορόσημα εκεί. Πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας Μίνσκ. Από αποτελεί προϋπόθεση. Θα πρέπει να έχουμε κοινή θέση απέναντι στις κυρώσεις και να είμαστε και ενωμένοι και βεβαίως και ε, τακτική διαβούλευση ώστε να, να μην στρεβλώνει το ανταγωνισμό. Όσοι από εσάς έχετε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζετε ότι υπάρχει πολύ έντονη δικοματική υποστήριξη για τις κυρώσεις σε δύο τομείς που εμείς παρακολουθούμε, τουλάχιστον από τη δική μου σκοπιά είμαστε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ο αγωγός Nord Stream 2, πολλές χώρες μέλη της Ένωσης, όχι όλες, η επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου είναι αντίθετη με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί μάλιστα να υποσκάψει και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενέργειας και μπορεί να βλάψει και την οικονομική βιωσιμότητα της Ουκρανίας καθώς και την ε, ε, ασφάλεια ενέργειας. Και αυτό το παρακολουθούμε λοιπόν. Και τέλος παρακολουθούμε σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση προμηθευτών ενέργειας την ε, υπόθεση ανταγωνισμού κατά της Γκασπρόμ. Η, η Ρωσία μπορεί και θα πρέπει να είναι ένας από τους προμηθευτές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να παίζει παιχνίδι με ισότιμου όρου ανταγωνισμού. Ορισμένε χώρε μέλη τη Ένωση έχουν εκφράσει ανησυχίε για τι προτινόμενε ε, ρυθμίσει, την προτινόμενη δηλαδή ε, εξοδικαστική ρύθμιση με την Gazprom. Αλλά θα δούμε που θα πάει αυτό το πράγμα. Πολύ σύντομα τώρα για, τις, για τους νέους κανονισμούς για τις αεροπορικές μεταφορές. Δεν έχω τις σχετικές πληροφορίες, βέβαια τα γνωρίζουμε εδώ και κάποιες μέρες την το αίτημα ορισμένες αεροπορικές γραμμές που ξεκινούν από ορισμένα αεροδρόμια, κυρίω ε, τη Μέση Μέσης Ανατολής. Απαιτούν μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές να πηγαίνουν στο αμπάρι του αεροσκάφους και να μην μπαίνουν μέσα στο, ε, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιβάτες εντός του αεροσκάφους. Αυτό είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε και συμφωνούμε και πολιτικά σε όλη την Ευρώπη αλλά και με τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή. Να πω λίγα λόγια. Σας ευχαριστώ που μου προσφέρετε νερό. Να έρθω με λίγα λόγια στο Μεξικό. Συμφωνώ. Η TPP, η ακύρωση της συμφωνίας TPP της ε, εταιρικής σχέσης του ειρηνικού ήταν κάπως μια έκπληξη ε, πρόκειται για μια συμφωνία η οποία φροντίζει για ανάπτυξη, όπως θεωρούν πολλοί, και μας επιτρέπει να στοχεύσουμε στη δημιουργία ενός συστήματος βασισμένου σε κανόνες. Η TPP μέχρι τώρα ήταν, ήταν ε, το απόλυτο στάνταρτ, το απόλυτο πρότυπο. Δεν συμφωνώ ότι είναι νεκρή η TPP. Ε, η TTIP, συγγνώμη, η TTIP δεν είναι νεκρή. Η άλλη συμφωνία δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει, γνωρίζω, μεγάλη υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ της TTIP και υπέρ της δημιουργίας ε, ανάπτυξης και απασχόλησης. Αλλά και στο Αμερικανικό Κογκρέσο υπάρχει μεγάλη υποστήριξη και η νέα Αμερικανική κυβέρνηση επανεξετάζει τη στάση της. Μην μονούμε βεβαίως κάποιες πρακτικές σκέψεις και να δούμε λίγο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπήκε κάπω στο ψυγείο η TTIP ή στη χαμηλή φωτιά αν θέλετε. Πρώτα-πρώτα ήταν το τέλος της ε, Αμερικανικής κυβέρνησης υπό τον πρόεδρο Ομπάμα. Υπήρχαν εκλογές, υπήρχαν και αλλού εκλογές και θεωρήσαμε ότι λόγω των δυσχεριών με τις επικείμενες Ολλανδικές, Γαλλικές και Γερμανικές εκλογές ότι δεν ήταν το καλύτερο κλίμα για να συνεχιστούν εμπορικές διαπραγματεύσεις για τις οποίες μεγάλο μέρος του κοινού είχε πολύ διαφορετικές απόψεις. Ήταν ίσως ζήτημα επικοινωνιακό, ίσως είχε πολιτικό χαρακτήρα. Πάντως πολλές ομάδες της κοινωνίας έχουν εκφράσει μια δυσαρέσκεια και ένα φόβο απέναντι στο εμπόριο είναι μια πραγματικότητα. Είτε πρόκειται για εγκαταλειμμένε ε, πόλει όπου ορθούσε κάποτε η χαλιβουργία, είτε πρόκειται για άλλε κοινότητε σε άλλα μέρη του κόσμου, στι ΗΠΑ. Ε, ε, ε, υπάρχουν πολλέ αμφιβολίε. Επανεξετάζουμε την συμφωνία και θα πρέπει κανείς να παραμείνει αισιόδοξο, διότι πρόκειται για μια σχέση, δεν είναι καμία μικρή συμφωνία μεταξύ δυο μικρών χωρών θα ήταν μια συμφωνία ανάμεσα στους δύο μεγαλύτερους συνασπισμούς, μεγαλύτερους, ισχυρότερους, πλουσιότερους και οικονομικά ισχυρότερους συνασπισμούς του κόσμου. Να πω τώρα λίγα για Λατινική Αμερική και Μεξικό. Μία συμφωνία που εξετάζεται τώρα από την Αμερικανική κυβέρνηση είναι η ναύτα. Πολλά λέχθηκαν σχετικά με την ναύτα και την εκ νέου διαπραγμάτευσή της. Οφείλω να πω ε, ότι έχουμε μια συμφωνία, Άντοα και Μέξικο City, που έχουν αρχίσει να το κάνουν αυτό. Και οι λόγοι. Πρώτα αναφέρομαι στην έννοια ότι θα πρέπει να εξηγηθεί το εμπόριο και εμπορικές συμφωνίες καλύτερα. Να εξηγηθεί η παγκοσμιοποίηση καλύτερα. Να αντιληφθούμε ότι κάποιοι τομεί θα έχουν ένα κόστος. Από την άλλη μεριά, η ναύτα χρονολογείται το 1994. Δηλαδή πολλά χρόνια. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Μιλούμε για μια εποχή πριν από τα FE τηλέφωνα, τα smartphone, πριν από τα iPad και τις άλλες ταμπλέτες, πριν από τις ροές δεδομένων, πριν από το ίντερνετ των πραγμάτων, πριν από την ανάπτυξη της οικονομίας των υπηρεσιών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που έγιναν τόσο κυριάρχες. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν και θα γίνουν. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους διαπραγματευτές μας το Μεξικό συνδέεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο μέσω του εμπόριου και της γεωγραφίας αλλά και με πολιτιστικούς και οικογενειακούς δεσμούς αλλά και πέραν αυτού αν δείτε τι έχει επιτύχει η ναύτα δηλαδή μια πλατφόρμα παραγωγής όπου παράγονται προϊόντα εκατέρωθεν των συνόρων και μεταφέρονται από τη μια στην άλλη μεριά. Θα τα εξετάσουμε αυτά και θα εξετάσουμε και ένα άλλο θέμα που ε, αφορά τα σύνορα, τη μετανάστευση. Πρέπει να εξετάσουμε πράγματι τη μετανάστευση, το πώς γίνεται, ε, οι υποκείμενες συνθήκες. Οι Αμερικανοί βλέπουν αυτή τη διαδικασία της μετανάστευσης ως άτακτη και ασυντόνιστη. Και νομίζω ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ε, μελετά κάποιους μηχανισμούς για να, την, για να βάλει μια τάξη. Δεν έχουμε αρχίσει επισήμως επανεξέταση της ναύτα, αλλά θεωρώ ότι αυτό θα γίνει. Δεν μπορώ να σας μιλήσω για την Γεωργία και την ένταξή τη ε, στο ΝΑΤΟ ε, δεν είναι τη δική μου αρμοδιότητα. Υπάρχει άλλο πρέσβη που ασχολείται με αυτά, ο μόνιμο αντιπρόσωπο στο ΝΑΤΟ. Να σα ε, αφήσω τώρα με μια τελευταία σκέψη. Σκεπτόμαστε όλοι, είμαστε πολιτικά ζώα εντό εισαγωγικών και βεβαίω έχουμε και εθισμό με τι πηγέ πληροφοριών. Πολλές πληροφορίε, προέρχονται βέβαια και από το Λευκό Οίκο. Οι πολιτικοί όμω, όπω γνωρίζετε και εσεί εδώ νομοθέτε είστε, δεν αποφασίζονται τα πράγματα αυτά μονάχα ε, μονομερός από τον Λευκό Οίκο, ούτε από κάποιους συμβούλους, ούτε μόνο από κάποιους υπουργούς. Όταν εγώ αποφύτησα από το Πανεπιστήμιο, ε, γινόταν τότε μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ Τζορτ Σούλτς και Κάσπαρ Βάινμπεργκερ, για όσους από εσά τα θυμάστε, για ε, ζητήματα άμυνας και εξωτερικών. Ε, μετά ε, στην ε, δεκαετία του 2000 μεταξύ Υπουργού Άμυνας τότε Ράμσφελτ και εξωτερικών Πάουερς. Αυτά που βλέπω είναι ότι το Κογκρέσο συμμετέχει πολύ ενεργά, διαθέτει μεγάλη εμπειρία, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, άλλωστε και θεσμικό, στο εμπόριο, καθορίζει τα του εμπορίου, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ως θεματοφύλακας των συμφερόντων των επενδυτών, των καταναλωτών, των εξαγωγέων όπως γνωρίζετε έχουν διεξαχθεί και πολλές συζητήσεις για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στις Ηνωμένε Πολιτείε με πρόσωπηση και των γερουσιαστών μας και βουλευτών μας σε θέματα εμπορίου και βεβαίως και χρηματοδοτήσεις ε, από ευρωπαϊκές επενδύσεις αλλά και το αντίστροφο και ολόκληρη Ουάσιγκτον, φίλοι, σύμφωνοι, όλοι παίζουν ένα ρόλο και χαίρομαι πολύ για το που βλέπω πόσοι πολλοί από εσάς έρχεστε στις Ηνωμένε Πολιτείες, συνεργάζεστε με αξιωματούχους του Κογκρέσου, οι άνθρωποι αυτοί έρχονται μετά εδώ, γνωρίζουν τη Σάρα Μακέιν, πρόκειται να έρθει. Ε, είναι όλα αυτά τμήματα μιας έντονης συζήτησης που συνεχίζεται. Και ο Λευκός Οίκος δεν είναι διαφορετικός. Διαβουλεύεται τακτικά και με δημοκρατικούς και με ρεπουμπλικανούς. Έτσι νομίζω εξελίσσεται και αναπτύσσεται η πολιτική. Και θυμίζω και το ρητό του Winston Churchill. Οφείλει να είναι κανεί αισιόδοξο γιατί τίποτε άλλο δεν αποδίδει. Εγώ είμαι αισιόδοξο. Το Brussels Forum που δημιουργήθηκε από το γερμανικό Marshall Fund και σε αυτό συνέρχονται και πολλοί πρώην ε, Αμερικανοί αξιωματούχοι και βεβαίω πάρα πολλοί Ευρωπαίοι και είναι θέματα τα οποία εκεί μπορούν να συζητηθούν που μα απασχολούν όλου. Ε, ευχαριστώ. Αγαπητέ Άνταμ Σούμπ, ευχαριστώ πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω ότι ακούσατε κι εσείς πολλές και χρήσιμες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ που τις, απαντήσατε, απαντήσατε και μακροσκελώς είπατε και στο τέλος κάτι που μου φαίνεται σημαντικό, ότι χρειάζεται να συνομιλούμε σε όλα τα επίπεδα. Σας ενθαρρύνω και εγώ να προσκαλέσετε να έρθουν εδώ όσο γίνεται περισσότεροι ε, ε, Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο πάντοτε είναι καλόδεχτοι να προσέλθουν εδώ είτε στην αντιπροσωπεία μας για τις σχέσεις με τα Αμερικάνικα νομοθετικά σώματα, είτε εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών. Σας εύχομαι καλή τύχη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και σας ευχαριστώ και πάλι που ήλθατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι το σημείο 12 στην ημερήσια διάταξη. Ωραία, θα σας δώσω λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να καθίσετε, and you never complain. May I ask our guest speakers to... Παρακαλώ τους προσκεκλημένους ομιλητές να έρθουν να καθίσουν εδώ. Εδώ μαζί μου, στο βήμα. Right, ladies and gentlemen. Καλώς, κυρίες και κύριοι. 10 και 5. Περνάμε στο επόμενο σημείο μας, στην ημερήσια διάταξη, το σημείο 12. Πρόκειται για ακρόαση με θέμα σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λατινικής Αμερικής και Καραϊδικής. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στις 11 και 25 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτό το θέμα, γιατί πολλοί από εμά θέλουμε να πάμε και να συμμετάσχουμε στην επαιτειακή εκδήλωση για τα 60 έτη από την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης, που είναι στις 11 και 30. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους εδώ στην ακρόαση αυτή, η οποία λαμβάνει η χώρα στα πλαίσια μιας έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας του κυρίου Χαμπί Λόπες, που είναι εισηγητής για αυτό το θέμα. Ευρωπαϊκή Ένωση, Λατινική Αμερική, Καραϊβική, οι σχέσεις αυτές έχουν αρχίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι βέβαια σε διάφορα επίπεδα, με πολυμερείς μηχανισμούς, αλλά και μέσω της συνέλευσης Eurolat. Για πολλούς και καλούς λόγους η εταιρική σχέση αυτή είναι στρατηγική σημασίας. Έτσι καθορίζεται. Οι παγκόσμιες προκλήσεις που έχουμε με τις εξελίξεις στον ε, Ατλαντικό μας οδηγούν να θέλουμε να ενισχύσουμε την εταιρική αυτή σχέση. Μια τέτοια ε, σχέση βασίζεται σε κοινέ αρχές και αξίες και στην πολυμερή διάσταση. Πρόσφατα συζητήσαμε την κατάσταση στην Βενεζουέλα Ακολουθούμε επίσης, παρακολουθούμε στενά την ενευτική διαδικασία στην Κολομβία και πολύ σύντομα θα ψηφίσουμε τη νέα συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κούβα. Να μερικά παραδείγματα δηλαδή πρόσφατων ε, συζητήσεων που είχαμε εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Οι σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής καλύπτουν και άλλους τομείς Εξού και έχουμε τέσσερις εξέχοντες προσκεκλημένους σήμερα να μας τα παρουσιάσουν. Έχουμε την κυρία Ρεμπέκα Γκρίνσπαν πρώτα απ' όλα, που είναι Γενικός Γραμματέας της Ιβυροαμερικανικής Διάσκεψης. Στη Κωνσταντίνα είχε αναλάβει διάφορα υπουργικά καθήκοντα, είναι από εκεί. Η επόμενη, η κυρία Πάουλα Μαντέη. Έχουμε και τον Κρίστια Έφνη που είναι αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ήταν διευθυντής ε, ε, Βόρειας και Νότιας Αμερικής. Έχουμε και την κυρία Πάολα Μαντέι, που είναι, γενική που είναι εκτελεστικός διευθυντής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Λατινική Αμερική και ε, Καραϊβική, το σχετικό ίδρυμα. Και τέλος έχουμε την κυρία Άννα Γιούσο Πόσο, που είναι ερευνήτρια για θέματα Λατινικής Αμερικής στο κέντρο διεθνών υποθέσεων της Βαρκελόνης και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης. Καλώς ήρθατε λοιπόν, είναι τιμή που σας έχουμε εδώ. Ο κύριος Λέπλερ έχει πρώτα το λόγο και μετά άλλοι πυρογνώμονες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Πάντα χαίρομαι όταν έρχομαι εδώ και μπορώ να συζητήσω με φίλους τις σχέσεις μας με την Αμερικανική Ήπειρο. Όπως γνωρίζετε, είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ, εκτός από μένα, και την ε, είπα το εκπρόσωπο, την κυρία Μογκερίνη, η οποία επενδύει πάρα πολύ στις διατλαντικές ε, σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις, τις διαστάσεις. Για σήμερα λοιπόν, εξετάζουμε τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής. Έχουμε λοιπόν ένα καλό παράδειγμα το τι θέλησε να φτιάξει η ύπατη εκπρόσωπος μέσω της παγκόσμιας στρατηγικής. Πώς δηλαδή θέλουμε να προωθήσουμε τη σχέση μας με τους εταίρους μας ανά το κόσμο. Θέλω από αυτού να ευχαριστήσω επίσης και τον ε, κύριο Χαμπιλόπες για την ε, πρωτοβουλία που ανέλαβε, για την έκθεση αυτή πρωτοβουλίας. Οι χώρες Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής μπορεί γεωγραφικά να βρίσκονται μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτιστικά όμως, διαρθρωτικά και πολιτικά βρίσκονται πολύ κοντά μας. Αυτή είναι η άλλη διάσταση των ε, διατρατικών μας ε, σχέσεων που συχνά ξεχνάμε ή υποτιμούμε. Ότι είμαστε συμπληρωματικοί. Η σχέση αυτή είναι συμπληρωματική σε σχέση με τη σχέση μας με τη Βόρεια Αμερική και εξίσου ισχυρή. Και η σχέση αυτή εκφράζεται όχι μόνο μέσω κοινών αξιών, κοινή ιστορίας, κοινών γλωσσών, αλλά εκφράζεται και στην πράξη πολύ ξεκάθαρα μέσω του τρόπου που αντιμετωπίζουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις και μέσω του πώς συνεργαζόμαστε σε διεθνές επίπεδο. Το είδαμε αυτό στις διαπραγματεύσεις που έγιναν για την κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα. Το είδαμε επίσης και στην προετοιμασία των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030. Το είδαμε στην ειδική συνέλευση επίσης που έγινε για τα ναρκωτικά. Και την προηγούμενη εβδομάδα, προκειμένου να δοθεί συνέχεια στην ετήσια διάσκεψη του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά. Στην Βιέννη, η Αμερικανική συμμετοχή των ε, χωρών αυτών, δηλαδή Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, ήταν πάρα πολύ αισθητή. Δεύτερον, έχουμε πολύ ισχυρέ οικονομικές σχέσεις μέσω εμπορικών επενδύσεων, συνεργασίας σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και όχι μόνο, ανάλογα με τον εταίρο μας. Και τρίτον, έχουμε κοινά συμφέροντα, προκειμένου να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε κοινέ ε, προκλήσεις που μας έχουν επηρεάσει και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Οργανωμένο έγκλημα, δημόσια ασφάλεια και διάφορα άλλα ζητήματα επίσης για τα οποία πρέπει να συνεργαστούμε για να τα λύσουμε. Και θα πρέπει ίσως να προσθέσω εδώ και μια τέταρτη διάσταση που είναι οι στενές σχέσεις μεταξύ των κοινωνιών μας, των ε, ανθρώπων, των, της κοινωνίας των πολιτών εκατέρωθεν του επιχειρηματικού κόσμου επίσης, των φοιτητών, των ερευνητών που έχουν ε, ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους. Πολύ σύντομα λοιπόν θα αναφερθώ τώρα σε τρεις τομείς όπου κατά το παρελθόν και τώρα συνεργαζόμαστε στενά. Κολομβία και ειρηνευτική διαδικασία είναι το ένα. Ο δεύτερος τομέας είναι η επέκταση και η ευάθυνση των συμφωνιών σύνδεσης που έχουμε με τις χώρες αυτές και το τρίτο είναι η κλιματική αλλαγή. Για την Κολομβία. Αποτελεί ένα από τα καλύτερα παραδείγματα που έχουμε για μια πλήρη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση διαχείρισης μετά από πρόσκληση των ε, αρχών της Κολομβίας και του Πρόεδρου μπορέσαμε και είπα πατή πρόσωπος και ειδικό ε, απεσταλμένος να στηρίξουμε συντονισμένα την ειρηνευτική αυτή διαδικασία και τεχνικά και οικονομικά και πολιτικά. Τώρα υπάρχει ένα καταπίστευμα ευρωπαϊκό, ένα trust fund, το οποίο, στο οποίο συμμετέχουν πολλές χώρες μέλη της Ευρώπης για να δείξουν ακριβώς την στήριξή του στη διαδικασία αυτή. Και όταν ε, ξεκίνησαν οι διαδικασίες της πολυμερούς εμπερικής ε, σχέσης, φάνηκε, ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία προκειμένου να συμμετέχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Κολομβίας. Υπήρχε δηλαδή μια νέα ευκαιρία για μια ευημερούσα και ειρηνική Κολομβία. Οι προκλήσεις βέβαια πολλές τουλάχιστον παραμένουν για το μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε έντονα τη στήριξή μας στην οικονομική, κοινωνική ζωή, ε, να δούμε τι θα γίνει με τους ΦΑΡ και πώς θα ενταχθούν στην κοινωνία, να διατηρηθεί η στήριξη του κόσμου στην ειρηνευτική διαδικασία επίσης στα πλαίσια των επόμενων εκλογών που θα γίνουν εκεί. Οι γειτονικέ χώρες, από την άλλη πλευρά, πρέπει και αυτές να συνεισφέρουν, να βρούνε το δικό δικό τους ρυθμό στήριξης, Βενεζουέλα για παράδειγμα, που πρέπει και εκεί να επανέλθει σταθερότητα και τα δημοκρατικά διαπιστευτήρια κατά κάποιο τρόπο, ώστε να υπάρξει διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Θέλω να ευχαριστήσω, επί τη ευκαιρία αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξή του στις δικές μας προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να διευκολύνουμε και να προωθήσουμε τον διάλογο αυτό στη Βενεζουέλα. Έρχομαι τώρα στις συμφωνίες σύνδεσης. Έχουμε μεγάλο δίκτυο σε ολόκληρη την Αμερικανική Ήπειρο και έχουμε δύο διαπραγματεύσεις αυτή την εποχή. Το ένα είναι για την αναβέθμιση της επιτυχούς συμφωνίας που έχουμε με το Μεξικό, είναι η συνολική συμφωνία αυτή. 15 ετών έγινε και θέλουμε να αντικατοπτρίζει τη σημερινή πραγματικότητα του Μεξικού και ευνόμαστε και από άλλε αντίστοιχε συμφωνίε όπω είναι η ΣΕΤΑ με τον Καναδά για να ενισχύσουμε τη συμφωνία αυτή. Επίσης έχουμε διαπραγματεύσεις και στα πλαίσια της Μέρκοσουρ για συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τεράστιο δυναμικό αυτές οι δύο συμφωνίες μαζί, Μέρκοσουρ ή μάλλον να το πω αλλιώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δούμε συνολικά το εμπόριο με τη Λατινική Αμερική και την Καραβική, 40% είναι ε, η Mercosur και 25% το Μεξικό. Δηλαδή τα δύο τρίτα των εμπορικών μας συναλλαγών καλύπτονται από αυτή τη συμφωνία. Καταλαβαίνετε τι δυνατότητες υπάρχουν. Και στο μέλλον οι επενδύσει θα είναι πιο σημαντικέ ακόμα. Αλλά οι συμφωνίε αυτέ δεν είναι μόνο εμπορικέ, πρόκειται και μια γενικότερη συνεργασία σε πολλού τομεί. Διάλογο, ευκαιρίε συνεργασία υπέρ των κοινωνιών μας ή ακόμα και σε περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο. Και για τους ίδιους λόγους αναβαθμίζουμε και την συμφωνία με την Χιλή. Και πρόσφατα έχουμε καλύψει τις, ε, τη συμφωνία με την Κούβα και ανθανένουμε τις χώρες μέλη να κυρώσουν την Περιφερειακή Συμφωνία Συνδύσης με την Κεντρική Αμερική. Αν πετύχουμε με τη Μερκοσούρ, με τις διαπραγματεύσεις αυτές, τότε θα έχουμε μια πλήρη επενδυτική και εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Λατινική Αμερική. Περισσότερο από ό,τι με οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο. Θα έχουμε τρεις εμπορικές ε, συμφωνίες που θα έχουμε προσφέρει στις χώρες αυτές, εκτός από την Κούβα, την Βολιβία και τη Βενεζουέλα. Κούβα στις διαπραγματεύσεις είπε η Κούβα ότι δεν ήθελε τέτοια συμφωνία ελεύθερου μπορείου, το σεβόμαστε. Η Βολιβία έχει έτσι κι αλλιώς ελεύθερη πρόσβαση επειδή πρόκειται για αναπτυσσόμενη χώρα και η Βενεζουέλα επειδή έχει άλλα ζητήματα που πρέπει να λύσει πριν φτάσει στο σημείο να μπορεί να πει σε διαπραγματεύσεις για τέτοια συμφωνία. Οι σχέσεις μας όμως είναι στενές και έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα συζητάμε αυτά τα θέματα. Και έρχομαι στο τρίτο που είναι η κλιματική αλλαγή. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία. Την είχαμε πριν εν ώψη τη Συμφωνία των Παρισίων και τώρα όσον αφορά την υλοποίησή τη. Και χαιρετίζουμε τι προσπάθειε που έχουν γίνει από την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική προκειμένου να υλοποιήσουν τη συμφωνία αυτή. Η Νικαράγουα δυστυχώ μένει εκτό γιατί αποφάσισε να μην υπογράψει τη συμφωνία κόπο των Παρισιών και ελπίζουμε ότι κάποια μέρα οι φίλοι τους θα τους ενθαρρύνουν και οι γείτονέ του να το κάνουν. Στο μεταξύ, πάνω από 20% της ε, χρηματοδότησής μας για τη συνεργασία την αφιερώνουμε στην κλιματική αλλαγή, να αντιμετωπιστεί δηλαδή αυτή η πρόκληση. Ξέρω ότι δεν έχω χρόνο, οπότε θα συμπληρώσω λέγοντας ότι με αυτά τα τρία παραδείγματα μπόρεσα να υπογραμμίσω πόσο καλά συνεργαζόμαστε στον τομέα ε, των πολιτικό, της ασφάλειας, πώς συνεργαζόμαστε με τις αρχές της Κολομβίας, πώς μπορούμε στον οικονομικό τομέα να συνεργαστούμε και να διευρύνουμε την εμπορική μας ατζέντα πέρα, από τις εμπορικές επενδύσεις και πώς πολυμερώς δουλεύουμε πάνω σε θέματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν και τα ναρκωτικά και άλλα. Στο τέλος της χρονιάς, τον Οκτώβριο, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη διάσκεψη που θα γίνει στο Ελ Σαλβαδόρ. Και ελπίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε μία επισκόπηση και να προγραμματίσουμε τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και στην δεύτερο. Η κυρία Ρεβέκα Γκρινσπάν είναι η επόμενη που έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που με επιτρέπετε να έρθω εδώ στην Επιτροπή αυτή. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Χάμπι Λόπες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας δίνετε την ευκαιρία αυτή. Αρχίζω λέγοντας, όπως το είπε και ο Κρίστιαν πολύ καλά, ότι Αυτές τις ε, μέρες είχαμε επαφές με τις αρχές Λατινική Αμερική και την Ευρώπη και κατάλαβα κι εγώ, ναι με καταλαβαίνετε εντάξει, και διαπίστωσα κι εγώ πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για την ενίσχυση των σχέσεων στα πλαίσια ε, τα σημερινά. Και Έχω την πεποίθηση ότι πρόκειται για μια στιγμή όπου προσφέρονται τεράστιες ευκαιρίες συνεργασίας ανάμεσα στη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη. Πριν από λίγο καιρό συναντήθηκα με την Φρεντερίκα Μογκερίνη, την είπα την εκπρόσωπο, σε μια συνάντηση που είχαμε και εκείνη επανέλαβε ότι οι σχέσεις είναι στενές και ιδιαίτερα ε, παραγωγικές και ότι αποτελεί πολύ συγκεκριμένο σημείο στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το είπε και ο προλαλής σας. Όντω είναι στρατηγική σημασία σε σχέση αυτή. Δεν πρόκειται μόνο για κάτι πρακτικό, είναι στρατηγικής σημασίας, όπως το επιβεβαίωσε και ο κύριος Σταγιάννη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόσφατα. Η σχέση αυτή φυσικά και εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια είναι σήμερα μια σχέση πολύ πιο συμμετρική και οριζόντια από ό,τι ήταν κατά το παρελθόν. Αλλά εξακολουθεί να βασίζεται, όπως το είπε επικεφαλής του πάνελ, σε κοινέ αξίες. Στην πολυμερή διάσταση, στη συνεργασία, στο διάλογο, στην βιώσιμη ανάπτυξη και στην ειρήνη. Αυτές οι αρχές αποτελούν τη βάση των σχέσεών μας με την Ευρώπη. Και όπως το έλεγε και ο Κρίστιαν πριν, η Λατινική Αμερική ήταν πάντα ένας πολύ βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως για να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη και να καταπολεμηθεί κλιματική αλλαγή. Αυτή η συμμαχία ανάμεσα στην Ευρώπη και την Λατινική Αμερική επέτρεψε να πετύχουμε φιλόδοξους στόχους στο διεθνές πλαίσιο. Οπότε, συμφωνούμε με την άποψη αυτή και πιστεύουμε και εμείς ότι η Λατινική Αμερική αποτελεί ένα σημαντικό εταίρο και όσον αφορά την ανταλλαγή αγαθών, αλλά και όσον αφορά την αντιμετώπιση παγκοσμίων προκλήσεων. Τώρα επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω κάποιο προβληματισμό για το τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Πρώτα απ' όλα υπήρξε πολύ σημαντική ανάπτυξη στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στις αρχές του αιώνα αυτού. Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια έχουμε ε, μια μεγάλη επέκταση στις τιμές των, ε, του διεθνούς εμπορίου των πρώτων υλών. Τεράστια ανάπτυξη. Κάτι το οποίο οδήγησε σε καλύτερη μακροοικονομική κατάσταση και μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Έτσι πήραμε το μάθημα της δεκαετίας του 80 και το μάθαμε και γι' αυτό καταλάβαμε τι έπρεπε να κάνουμε μετά από την κρίση που ξεκίνησε με την ιστορία της Lehman Brothers. Για πρώτη φορά λοιπόν αυτή η οικονομική ανάπτυξη και αυτό, αυτός ο οικονομικός δυναμισμός μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια στις χώρες μας. Καταφέραμε να συνδυάσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στην περιοχή, αλλά επιπλέον, αυτό το είχαμε κάνει και παλιότερα, αυτό όμως που επιπλέον κάναμε ήταν ότι μειώσαμε τις ανισότητες. Είναι μεγάλο επίτευγμα στην περιοχή. Γιατί παντού μειώθηκε η φτώχεια τα τελευταία χρόνια. Η μόνη περιοχή του κόσμου όμως όπου μειώθηκαν οι ανισότητες ήταν στην Λατινική Αμερική και την Καρυβική. 0,7% το χρόνο. Η ερώτηση λοιπόν είναι, αυτό οφείλεται μόνο στην οικονομική ανάπτυξη ή και στις δημόσιες πολιτικές που συνόδευσαν την οικονομική αυτή ανάπτυξη. Και η απάντηση, σύμφωνα με τις αναλύσεις και τις έρευνες που έχουν γίνει, είναι ακριβώς ότι η οικονομική ανάπτυξη φυσικά και έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης στην αγορά εργασίας, στην απασχόληση, αλλά βοήθησε και την εκπαίδευση. Αν δεν υπήρχε η σωστή εκπαίδευση, ο κόσμος που θα μπορούσε να πάει στην αγορά εργασίας δεν θα μπορούσε να αποφεληθεί από καλές δυνατότητες απασχόλησης. Άρα λοιπόν η μείωση των ανισοτήτων οφείλεται στην αύξηση της απασχόλησης αλλά και στις κοινωνικές πολιτικές. Ποιες κοινωνικές πολιτικές? Την μεταφορά πόρων αλλά κυρίως την εκπαίδευση και την υγεία. Ο αγώνας που δώσαμε για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και υπέρ των αυτόχθανών πληθυσμών. Το πρόβλημα των ανισοτήτων αντιμετωπίστηκε οριζόντια και αποτέλεσε μέρος της πολιτικής των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Οπότε αυξήσαμε την απασχόληση, αυξήθηκε ο ελάχιστος μισθός και βελτιώθηκε το θέμα της ισότητας. Όμως, τώρα παραμένουν κάποιες εκκρεμότητες, γιατί δεν λύθηκαν όλα. Οπότε, ναι, ε, στην αρχή ανέβηκε η τιμή των πρώτων μετά έπεσε και τώρα λοιπόν πρέπει να πληρώσουμε το λογαριασμό. Ποια είναι η χιλίος πτέρνα το τι δεν κάναμε στο διεθνές πλαίσιο. Ήτανε ότι δεν διαφοροποίησαμε επαρκώς τον παραγωγικό μηχανισμό. Δηλαδή βασιστήκαμε στα αγροτικά προϊόντα για τις εξαγωγές μας και είχαμε μια παραγωγικότητα που λίγο ανέβηκε τα τελευταία χρόνια. Η Ασία αύξησε την παραγωγικότητά της πολύ περισσότερο από ό,τι το έκανε η Λατινική Αμερική. Συνεπώς είχαμε μια επανάσταση κατά κάποιο τρόπο στην ε, παραγωγικότητα και χρειαζόμαστε τώρα πολιτικές παραγωγικής ανάπτυξης που να μας επιτρέψουν περισσότερες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, στη γνώση και καταπολέμηση των άτυπων μορφών παραγωγής. Και όλα αυτά στα πλαίσια βέβαια μιας νέας διεθνούς σκηνής. Υποδομές τώρα. Οι υποδομές είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο για να συμμετέχουμε στο διεθνές εμπόριο αλλά και στην περιφερειακή ολοκλήρωση. Ένα άλλο θέμα ήταν η κοινωνική προστασία που δεν έγινε συνολικά. Εξακολουθούν κάποιοι άνθρωποι να βρίσκονται κάτω από το όριο φτώχεια στις χώρες μας και να υποφέρουν από χαμηλή οικονομική ανάπτυξη για την έμενα, αλλάξαμε την κοινωνική μας δομή, αλλά το 1 τρίτο του πληθυσμού μας είναι μέσα τάξη, αλλά υπάρχουν και ένα τρίτο που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας και ένα τρίτο το οποίο βρίσκεται στο ευάλωτο κομμάτι ανάμεσα στα δύο. Γι' αυτό χρειάζονται πιο οικουμενικές ε, δομές κοινωνικής προστασίας. Όπως έλεγε και ο Κρίστιαν, έρχεται εδώ και το θέμα της ανασφάλειας. Ε, η βία και η αστικοποίηση. Λατινική Αμερική είναι η περιοχή του κόσμου που το 80% του πληθυσμού ζει σε πόλεις, στην πόλη. Και αυτό έχει να κάνει και με τόσα είπα πριν. Συνεπώς, αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερη ολοκλήρωση με την Ευρώπη, αλλά και μέσα στην ίδια τη Λατινική Αμερική. Και γι' αυτό, Κριστιαν, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες πριν, ότι πρέπει να ενημερωθούν οι συμφωνίες με τη Χιλή και το Μεξικό και να υπάρξει πολιτικός διάλογος με την Κούβα. Αυτά είναι στοιχεία πολύ σημαντικά για να πετύχουμε αυτή τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση που θέλουμε όχι μόνο με την Ευρώπη, αλλά και μέσα στην ίδια την περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής, όπως είπα. Γιατί αν υπάρχει συμφωνία με τη Σούρ είναι γιατί καταφέραμε με τη Συμφωνία σύνδεση με την Ευρώπη να έχουμε και μεταξύ μας καλύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση. Εκεί είμαστε σε ένα στάδιο πια που μπορούμε να μιλάμε για προέλευση προϊόντων, μπορούμε να μιλήσουμε για περισσότερη εναρμόνιση των συμφωνιών σύνδεσης που έχουμε με την Ευρώπη. Αυτό βοηθάει την ολοκλήρωση του Λατινική Αμερική. Και θα τελειώσω με το εξής. Βρισκόμαστε σε μια πολύ λεπτή στιγμή για την περιοχή. Κρίσιμη. Έχουμε ε, ένα μεγάλο ποσό του πληθυσμού που είναι νέοι, που ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Αν δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, αμφισβητείτε το κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί η Λατινική Αμερική. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συμβιβάσουμε τις προσδοκίες του κόσμου με την ικανότητα του οικονομικού και πολιτικού συστήματος. Και υπάρχουν και τα προβλήματα διαφθοράς, τα οποία παρουσιάστηκαν και έγιναν ε, εμφανή τα τελευταία χρόνια, παρόλο που σήμερα γνωρίζουμε τα ονόματα των ε, ε, δικαστών, όχι των στρατηγών. Παλιά συνέβαινε το αντίθετο. Οπότε αυτό δείχνει τη θεσμική αλλαγή που έχει επέλθει στη Λατινική Αμερική χάρη στη συνεργασία με την Ευρώπη σε τομείς, τεχνολογία, επιστήμες, κλιματική αλλαγή. Όντως πετύχαμε πολλά. Η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική έχουν κοινούς στόχους σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Για 10 λεπτά η κυρία Μαντέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή να έρθω και να μιλήσω στην Επιτροπή σας μαζί με άλλους πρωταγωνιστές των σχέσεων της Ευρώπης με τη Λατινική Αμερική και την Καρεβική. Πολύ σύντομα θα σας παρουσιάσω το Ίδρυμά μας, το ΕΟΛΑΚ. Είμαι εκτελεστικός διευθυντής. Το Ίδρυμα αυτό δημιουργήθηκε από τις 33 χώρες μέλη της ε, ΣΕΛΑΚ και τις 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια. Και λειτουργεί από το 2011 στο Αμβούργο, που είναι η έδρα μας. Τα μέλη του Ιδρύματος έχουν αναθέσει στο Ίδρυμα να ενισχύσει την ε, στρατηγική σχέση στην περιοχή να ενισχύσει τις κοινωνίες των πολιτών και να προωθήσει την προβολή του ίδιου του Ιδρύματος. Ο πιο σύντομος ορισμός που θα μπορούσα να δώσω για το έργο του Ιδρύματος έρχεται από την ίδια την είπα το εκπρόσωπο Μογκερίνη, η οποία είπε ότι τα καθήκοντα του Ιδρύματος είναι να προβάλλει στο μέλλον τις ιστορικές και παραδοσιακές σχέσεις των δύο πλευρών την ε, υπουργική συνάντηση της ΕΛΑΚ που έλαβε χώρα στο Σάντο Ντομίνγκο τέλη Οκτωβρίου υπογράφηκε η ιδρυτική πράξη του Ιδρύματος για τη συνεργασία του με άλλους διεθνείς οργανισμούς και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε μέχρι τα τέλη της χρονιάς να έχουμε πετύχει τις 16 κυρώσεις που χρειάζονται. μεταξύ άλλων και εκείνη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό βέβαια σας το λέω ότι η Επιτροπή σας μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Τώρα είμαστε σε μια στιγμή όπου οι πολίτες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα εσωτερικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις συγκρούσεις κοντά στην Ευρώπη, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τη σημασία που έχει η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Η πρωτοβουλία λοιπόν που αναλάβατε για έκθεση δύο πρωτοβουλίες για τις σχέσεις αυτές είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Και στις δύο περιοχές και σε διαφορετικό επίπεδο βέβαια, δημιουργείται η αντίληψη ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα business as usual, αλλά ότι χρειάζεται να δοθεί νεόθεση στη σχέση αυτή, μια που έχουμε κοινά συμφέροντα και πρέπει να υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες υπέρ των πολιτών. στη σημερινή τη σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να υπογραμμίσει τον ρόλο της ΣΕΛΑΚ ως στρατηγικό εταίρο υπέρ μιας βιώσιμης ανάπτυξης, υπέρ ενός ισότιμου και δίκαιου εμπορίου και υπέρ της, πολυ... της πολλαπλής διάστασης, της πολυμερούς διάστασης. Οι δύο περιοχές ε, έχουν πολλές κοινέ αξίες και προτεραιότητες: Βιώσιμη ανάπτυξη, προώθηση της κοινωνίας των πολιτών χωρίς ε, αποκλεισμούς, οικονομική ανάπτυξη. Ήμασταν πάντα στην πρώτη γραμμή για διάφορες ε, συμφωνίες. Αναφέρθηκε πριν ο ρόλος των δύο περιοχών προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και η Συμφωνία των Παρισίων μπορούμε να μιλήσουμε και για τη συμφωνία μεταξύ των δύο περιοχών που όντως βοήθησε σε επίπεδο του ΙΕ να υπάρξει συμφωνία για τον περιορισμό των λαφρών όπλων. Μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε σε λύσεις, να αποφεύγουμε συγκρούσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε να λέμε ότι οι δύο αυτές περιοχές του κόσμου είναι δύο περιοχές που στη βάση της συνεργασίας τους έχουν την ενίσχυση της ειρήνης. Και αυτό είναι μοναδικό σε διεθνές επίπεδο. Και δεν θέλω να παραλείψω να αναφερθώ και στους μετανάστες. Είτε τους Ευρωπαίους στην Λατινική Αμερική, που βέβαια είναι δεύτερης, τρίτης γενιάς, αλλά υπάρχουν και νέοι, και από την άλλη υπάρχουν και οι μετανάστες από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική στην Ευρώπη. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε ε, τις σχέσεις λοιπόν μεταξύ των δύο πλευρών, ακριβώς να τις δούμε και από την οπτική γωνία των μεταναστών αυτών. Τώρα, υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρήσουμε δεδομένες τις αξίες που συμμεριζόμαστε και να μην συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας ενίσχυσης των σχέσεων αυτών κάτι το οποίο μπορεί να μας ε, βοηθήσει γιατί έχουμε να μάθουμε ένας από την εμπειρία του άλλου. Μπορεί να σε βεί όπως συμβαίνει πολλές φορές ε, στην ε, ταινία του Μπέρκμαν στο ζευγάρι που κρύβανε τα προβλήματά τους κάτω από το χαλί και τελικά φτάσανε να αρχίσουν να ψάχνουν άλλο σύντροφο για να νεώσουν την σχέση τους. Αυτό κινδυνεύει να συμβεί και με τις Δικέ μας περιοχές. Αλλά για να μην συμβεί πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί τα σημερινά προβλήματα, να έχουμε καρποφόρο διάλογο που να λαμβάνει υπόψη τους όλες τις πτυχές. Και ακριβώς εκεί είναι που το δικό μας το Ίδρυμα μπορεί να βοηθήσει. Οι δικές μας δραστηριότητες ακριβώς διευκολύνουν τον διάλογο. Όχι μόνο μεταξύ εκπροσώπων κυβερνήσεων, αλλά χρησιμοποιώντας και την ζωντανή δύναμη των κοινωνιών μας. Στα πέντε χρόνια που λειτουργούμε, προωθήσαμε τη συνεργασία μεταξύ ιδρυτημάτων ανώτατης εκπαίδευσης και φροντίσαμε να υπάρξει προσέγγιση και στον τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Προσπαθήσαμε να βρούμε και κοινέ λύσεις για την κοινωνική ευθύνη των εταιριών. Για να λύνουμε διλήμματα που υπάρχουν στις κοινωνίες μας, πρέπει να βασιζόμαστε σε κοινή γνώση μεταξύ των δύο ε, περιοχών. Σε αυτό δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε ένα σύνολο προγραμμάτων και από τις δύο πλευρές το ευρωσοσιάλ, ευρωκλίμα, ε, ορίζοντας 2020, που πολλά life κτλ. Προγράμματα τα οποία άνοιξαν το δρόμο που προωθεί την οριζόντια συνεργασία με συμμετοχή παραγόντων των κοινωνιών μας. Είμαι σίγουρη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα βρισκόταν στην πρώτη γραμμή προκειμένου να στηρίξει προγράμματα όπως το Έρασμος με συμμετοχή τρίτων χωρών. Και αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα προγράμματος που προσεγγίζει τις ζωντανές δυνάμεις των κοινωνιών μας, τις φέρνει πιο κοντά. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί ένα εκπληκτικό εργαλείο υπέρ της συνεργασίας. Θα συνεχίσω στα αγγλικά που επίσης είναι και γλώσσα εργασίας του Ιδρύματος μαζί με τα Ισπανικά. Θα ήθελα... Αυτό μας δείχνει και την ποικιλομορφία που υπάρχει και σε γλωσσικό επίπεδο των περιοχών μας. Δείχνει και πόσο σημαντικό είναι σε αυτή την εταιρική σχέση να συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέλη και εκείνου που λόγω μεγέθους ιστορίας, τοποθεσίας και πολιτισμού είχαν ενταχθεί λιγότερο στις παραδοσιακές συνομιλίες και επαφές των δύο περιοχών του κόσμου κατά το παρελθόν. Γι' αυτό το λόγο επίσης το Ίδρυμα έχει καταρτήσει ειδικά προγράμματα που απευθύνονται από τις χώρες Βίζεγκράτ προς την Καραϊβική, προς τις Βαλτικές χώρες, ούτως ώστε να ευνοήσουμε πληρέστερη διάδραση. Η παρουσίασή μου δεν θα μπορούσε να είναι πλήρης αν δεν αναφερόταν πέρα από τις ευκαιρίες και στα προβλήματα που επηρεάζουν τις περιοχές αυτές και χρειάζεται αμοιβαία συνεργασία για τη λύση των προβλημάτων. Θα περιγράψω τρία θέματα, ανισότητα, φτώχεια, ο ευάλωτος χαρακτήρας της δημοκρατίας για τη φτώχεια και την ανισότητα, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, Ήδη αναφέρθηκε εκτενώς αυτά. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι στα υποθέντα. Πράγματι, βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια και μια διαδικασία για τιμή των ισοτήτων, αλλά έχει αποτελματωθεί και ίσως να έχουμε και μια επιδείνωση της καταστάσεως. Χρειαζόμαστε περισσότερη ολοκλήρωση. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η πρόθεση των συμφωνιών σύνδεσης και να εφαρμόζονται αυτές και πρέπει να συνεχίσουμε την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγών εμπειριών, προγραμμάτων οριζοντίου συνεργασίας ε, για κοινωνική ένταξη και βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα, ο ευάλωτος χαρακτήρας των δημοκρατιών και στις δύο περιοχές βλέπουμε ότι υπάρχει μια απογοήτευση όσον αφορά τη δημοκρατία. Μια απομάκρυνση. Και ξέρουμε, είναι συνέπεια των κοινωνικών συνοπιών, της οικονομικής κρίσεως, καταναγκαστικής ε, μετακίνησης πληθυσμών και βιών συγκρούσεων. Σαν ευρωπαϊκοί νομοθέτες που ενδιαφέρεστε τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και την Καρυβική, προσβλέπουμε σε εσάς μπορείτε να αναπτύξετε καινοτόμα μέσα για να ανταποκριθείτε στο αίτημα των πολιτών για τη δημιουργία πολιτικών συστημάτων και να συνεχίσετε εφαρμογή πολιτικών οι οποίες θα μπορούσαν να επιλύσουν τα διάφορα προβλήματα. Και να μειωθεί η απογοήτευση των δημοκρατικών θεσμών. Οι χώρες Ατρικής Αμερικής και Καραϊβικής βλέπουν σαν πρόβλημα το θέμα της ταξινόμησης όσον αφορά τα εισοδήματα των χωρών. Κλείνοντας για αυτή τη διαβάθμιση, πράγματι χρειάζεται αναβάθμιση της συνεργασίας. Αυτή η διαβάθμιση, αυτή καθεαυτή, υπήρξε επιτυχής να διακόπτεται η συνεργασία απότομα ίσως να έχει αρνητικές συνέπειες θα πρέπει να βρεθεί μια λύση γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Πόσολη, τελευταία εμπειρογνώμων για το ίδιο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να συμμετέχουμε. Ακούστηκαν ε, πολλά, δεν θα τα επαναλάβω, θα επικεντρωθώ σε όσα δεν ακούσαμε. Είναι αλήθεια ότι οι δεσμοί μεταξύ των δύο περιοχών και οι μακρές ε, σχέσεις αποτελούν ε, μια πολύ στέρεα βάση για να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και μια κόπωση, γι' αυτό και πρέπει να βρούμε μια νέα, ένα νέο δρόμο, μια νέα στρατηγική που θα ξαναδημιουργήσει αυτή τη σπίθα η οποία λείπει τα τελευταία χρόνια και έχει οδηγήσει στην κόπωση. Χρειαζόμαστε ευκαιρίες στους νέους στόχους που μπαίνουν διεθνώς και που απαιτούν τέτοιες σχέσεις στρατηγικής σημασίας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε διαφορετικού τύπου σχέσεις μεταξύ μας επιπλέον. Είπαμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε και τη σύγκρουση συμφερόντων που υπάρχει, γιατί δεν μπορούμε να τα κρύβουμε. Πρέπει να βρίσκουμε λύσεις σε τέτοιες περιπτώσεις, και να τις δούμε αυτές τις συγκρούσεις συμφερόντων σαν νέες ευκαιρίες εφόσον θα λυθούν. Δεν μιλήσαμε για τις σχέσεις οικονομικές κλπ. Είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη έχει μειώσει την παρουσία της στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να τα αναγνωρίσουμε αυτό. Ε, για διορθωτικούς λόγους μερικές φορές που θα παραμείνουν, για το γεγονός ότι υπάρχουν νέοι παράγοντες, ότι η Λατινική Αμερική και αυτή έχει στραφεί προς την Ασία για την ανάπτυξή της, αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη της η Ευρώπη. Συνεπώς η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει σε αυτά τα γεγονότα και να λάβει υπόψη της ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες εκείνες οι οποίες μας οδηγούν σε συνεργασία με άλλους εταίρους. Δύο άλλα θέματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για τη συνέχεια και στο οποίο πρέπει να ανταποκριθούμε διαφορετικά είναι το θέμα της έλλειψης συμμετριών. Η Ευρώπη με τη Λατινική Αμερική είχαν ασυμμετρικές σχέσεις εξαιτίας διαφορετικής ανάπτυξης διαφορετικού επίπεδου ανάπτυξη. Τώρα αυτό έχει αλλάξει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Οι ασυμμετρίες όμως παραμένουν και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις σχεσεις ευρωπη Ευρώπη-Λατινική Αμερική έχουν να κάνουν και με τις σχέσεις μέσα στην ίδια την Λατινική Αμερική, αλλά και μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Και εκεί υπάρχουν ασυμμετρίε. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα οδηγηθούμε ξαφνικά σε μια απόλυτη συμμετρία. Όχι, θα είναι μια σχετική συμμετρία, γιατί εξακολουθούμε να μην είμαστε ομοιογενείς. Και μάλιστα σήμερα ίσως, εντάξει, μπορεί λιγότερο από ό,τι κατά το παρελθόν, από την άλλη μεριά όμως υπάρχει περισσότερη αμφισβήτηση, υπάρχει μια πιο ισχυρή διάσταση περιφερειακή, ο ρόλος της περιφερειακής αυτής διάστασης έχει ενισχυθεί. Παρά τις κρίσεις από τις οποίες έχει περάσει, εξακολουθεί να είναι ένα βασικό στοιχείο των ε, σχέσεων των δύο περιοχών. Γιατί μετά από κάθε κρίση περάσαμε σε λύσεις. Τις ξεπεράσαμε δηλαδή αυτές τις κρίσεις κάθε φορά και κάθε φορά που γίνονται διαπραγματεύσεις για νέες συνθήκες, αυτή η διάσταση περιφερειακή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, έτσι ότι δημιουργείται δηλαδή μία περιφέρεια στη Λατινική Αμερική χωρίς κατακαιρματισμούς, πιο συνολική. Άρα πρέπει να είναι συμβατό το να υπάρχει διμερή σχέση αλλά συγχρόνως με την περιφερειακή διάσταση που υπάρχει στον κόσμο και που είναι τρόπος διακυβέρνησης. Αναφέρεται και στους αναπτυξιακούς στόχους και η Συμμαχία Ευρώπης Λατινικής Αμερικής περνάει μέσα και από την περιφερειακή αυτή διάσταση. Τώρα, οι σχέσεις μεταξύ μας έχουν πολύ ισχυρή θεσμική διάσταση. Εντάξει, είμαστε στρατηγικός εταίρος, όπως με τις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά η θεσμική διάσταση περιλαμβάνει την πολιτική διάσταση με υψηλού επίπεδου διάλογο που μας κάνει να καταλαβαίνόμαστε καλύτερα και να γνωριζόμαστε καλύτερα συζητιούνται τα κοινωνικά θέματα. Παλιά η κοινωνική συνοχή δεν ήταν κάτι πάνω στο οποίο συμφωνούσαμε. Τώρα ναι. Και οφείλεται στο διάλογο, στη διάσταση του διαλόγου. Επίσης, έχουμε και διάφορα εργαλεία συνεργασίας. Όμως, Ανάμεσα στις διάφορες πτυχές υπάρχουν ασυνέπειες που πρέπει να τις προσέξουμε. Έχουμε το πρόγραμμα δράσης της ΣΕΛΑΚ, έχουμε τα στρατηγικά σχέδια, έχουμε πολλά προγράμματα. Όλα αυτά όμως πρέπει να φροντίσουμε να είναι μεταξύ τους συμβατά και να συμπεριλαμβάνονται στην συνολική ατζέντα. στους στόχους, δηλαδή του 2030, κλιματική αλλαγή κλπ. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει τη, τους στόχους της διμερούς σχέσης να τους βάλουμε μέσα στα πλαίσια μιας πιο πολυμερούς σχέσης. Κάτι άλλο είναι ότι σήμερα υπάρχουν άπειροι φορείς στις σχέσεις αυτές δεν πρόκειται μόνο για σχέσεις μεταξύ χωρών, αλλά πρόκειται και για σχέσεις μεταξύ πανεπιστημίων, κέντρων, κοινωνία των πολιτών, επιχειρήσεων. Είναι μια πολυεπίπεδη διαπεριφερειακή σχέση. Αυτό είναι καλό, γιατί μας βοηθάει να έχουμε δίκτυα ανταλλαγών, αλλά μπορεί να αποδυναμώσει κάπως την προσπάθεια για τον προσανατολισμό. Υπάρχουν και δυναμίες στη σχέση. Μία από αυτές είναι η έλλειψη πολιτικών προτεραιοτήτων, ε, λείπουν δηλαδή πολιτικές προτεραιότητες σε σχέση με την Ευρώπη, στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Δεν τη θεωρούν προτεραιότητα. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε. Εγώ συμμετείχα σε μια μελέτη για τις σχέσεις Ανατολικής Ευρώπης με τη Λατινική Αμερική. Και είδαμε ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και καλύτερη γνώση που χτίζεται βέβαια σιγά σιγά, δεν μπορεί να θεωρηθεί κάτι δεδομένο. Οι αδυναμίες μας ποιε είναι. Τα συμμετρικά σοκ. Δεν ξέραμε και δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις. Δημιουργούνται και στο εσωτερικό των περιφερειών κρίσης. Εμείς πήραμε κάποια μαθήματα, μάθαμε, διορθώσαμε κάποια. Δεν ξέρω κατά πόσο και η Ευρώπη μπόρεσε να υποφεληθεί από τις δικές μας κρίσεις. Σε αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο αλλά πρέπει να δούμε πώς την διαπεριφερειακή αυτή σχέση και τους στόχους της, πώς μπορούμε να τους προσαρμόσουμε στο διεθνές πλαίσιο. Όντως πρέπει να ενημερώνονται οι συμφωνίες, να προσαρμόζονται βάσει των αναπτυξιακών στόχων. Υπάρχουν οι διαπραγματεύσει στην Τόχα, υπάρχουν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που δεν πρόκειται για μια συνεργασία, πρόκειται για ανάπτυξη και για τις δύο περιοχές. Έχουμε κοινούς στόχους. Φυσικά όχι τις ίδιες ευθύνες, γιατί οι δυνατότητες είναι διαφορετικές στην Ευρώπη και στην Λατινική Αμερική. Συνεπώς, τους στόχους αυτούς πρέπει να τους προωθήσουμε, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έχουμε διαφορετικές ευθύνες προκειμένου να τους φέρουμε σε πέρας και μέσα σε μια περιοχή στη Λατινική Αμερική, δηλαδή στην Ευρώπη, κάθε χώρα έχει διαφορετικές ευθύνε ανάλογα με τις ικανότητε τη. Είπαμε και για τις ανισότητες, που είναι κάτι το οποίο έρχεται και επανέρχεται και στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια η Λατινική Αμερική έχει κάνει τεράστια πρόοδο, αλλά το θέμα παραμένει στους ε, στόχους και της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης δεν είναι μόνο θέμα ανακατανομής. Πρέπει να αλλάξουν πολλά από τον τρόπο παραγωγής, διάφορα ρυθμιστικά πλαίσια για απασχόληση ποιότητας, κυκλική οικονομία και θα φέρω και ένα άλλο ζήτημα, τη ρομποτική και τι απασχόληση δημιουργείται με τη ρομποτική. Κοινωνία της γνώσης. Και κάτι ακόμα που θα βρίσκουμε μπροστά μας όλο και περισσότερο είναι οι δημογραφικές αλλαγές. Η Ευρώπη ξέρουμε τι εξελίξεις έχει στο δημογραφικό. Η Λατινική Αμερική επίσης είπαμε ότι είναι η περιοχή του κόσμου με περισσότερο αστικό πληθυσμό. Και για να ολοκληρώσω, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η συνοχή των πολιτικών. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στη συνεργασία μας, πρέπει να υπάρχει καλός συντονισμό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Λόπες, για ένα πεντάλεπτο για να ξεκινήσει η συζήτηση και μετά θα δώσουμε το λόγο σε συναδέλφους που έχουν ζητήσει. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους προσκεκλημένους μας. Και τη Ρεβέκα και τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, την Πάολα, ε, την Άννα όλους. Είναι πολύ καλό που μπορούμε να σας ακούσουμε έτσι από πρώτο χέρι για να ετοιμάσουμε τη δικιά μας έκθεση πρωτοβουλίας. Να ακούσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας. Εσάς που δουλεύετε πάνω στην περιοχή σε καθημερινή βάση. Θέλω να εξηγήσω λιγάκι γιατί αποφασίσαμε να αναλάβουμε την πρωτοβουλία της έκθεσης αυτής. Γιατί Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις και ποιο είναι το έργο μας τους τελευταίους 7 μήνες στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, αποφασίσαμε να κάνουμε την έκθεση αυτή πρωτοβουλία ακριβώς γιατί ε, θεωρήσαμε ότι η Λατινική Αμερική πρέπει να επανέλθει στην κοινοβουλευτική συζήτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει βοηθήσει τα τελευταία 7 χρόνια βέβαια σε αυτό. Το 2010 είχαμε την έκθεση Σαλαφράνκα που εργάστηκε πολύ για τις σχέσεις αυτές. Τα τελευταία όμως έξι χρόνια έγιναν πάρα πολλά, τόσο στη Λατινική Αμερική όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γίνονται και πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο ολόκληρο. Οπότε προφανώς και πρέπει να υπάρξει κάποια προσαρμογή των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ μας. Θέλαμε λοιπόν να στείλουμε το μήνυμα ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα οι σχέσεις μας με τη Λατινική Αμερική είναι στρατηγική σημασία. Γιατί τις, ε, την άποψή μας για τις διεθνείς ε, σχέσεις την ε, μοιραζόμαστε με τη Λατινική Αμερική περισσότερο από ό,τι με οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου. Το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, πώς θα προχωρήσουμε στην οικονομική ανάπτυξη. Με κανέναν άλλον δεν έχουμε τόσο κοινέ απόψει όσο έχουμε τη Λατινική Αμερική. Και το 2016 βέβαια μας οδήγησε σε ένα διαφορετικό κόσμο. Είχα μια διαφορετική διεθνή σκηνή Άρα τις προτεραιότητές μας πρέπει να τις επανακαθορίσουμε. Μια νέα προτεραιότητα για μας λοιπόν δίχως άλλο είναι η Λατινική Αμερική. Έχουμε κοινέ αξίες, κοινά συμφέροντα. Είμαστε μια κοινότητα αξιών, αρχών, συμφερόντων. Έχουμε και κοινού πολιτικούς στόχους πάνω στους οποίους έχουμε δουλέψει τα τελευταία χρόνια ανάπτυξη για όλους, κοινωνική ευαισθησία, κλιματική αλλαγή, ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, ε, ψηφιακέ αλλαγές. Έχουμε και κοινέ απειλές να αντιμετωπίσουμε με διαφορετική μορφή. Ασφάλεια, εμείς λόγω της τρομοκρατίας, η Λατινική Αμερική έχει να αντιμετωπίσει περισσότερο το οργανωμένο έγκλημα, ε, υπάρχουν ε, αδυναμίες όσον αφορά την κοινωνία που είναι μέρος της ιδιαίτερα ευάλωτο. Και έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θέλει να καλύψει πολιτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνίες δηλαδή όπως η Μερκοσούρ, η προσαρμογή των συμφωνιών μας με το Μεξικό και τη Χιλή, Κούβα. Όλοι αυτοί είναι στόχοι που έχουμε για τους επόμενους μήνες και χρόνια και γι' αυτό θέλαμε να στείλουμε το μήνυμα αυτό ότι υπάρχει αυτή η πολιτική κάλυψη από την πλευρά μας. Επίσης, στους επόμενους μήνες ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν και οι καταστάσεις. Μετά τη δικιά μας εργασία για την έκθεση αυτή, όπου θα συμμετάσχουν όλοι, στην συνέχεια θα έχουμε το φθινόπωρο μία διάσκεψη σε ΛΑΚ και το Σεπτέμβριο στο Σαλβαδόρ της Eurolat που είναι η συνέλευση εκείνη η οποία λειτουργεί καλύτερα από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει τα εργαλεία που χρειάζονται, τη διπλωματική διάσταση με μεγάλη ιστορία από πίσω. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σκεφτεί καλά τις σχέσεις που έχουμε με τη Λατινική Αμερική. Αν λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία τα βάλουμε μαζί, ξέρουμε ότι θα μπορέσουμε να επανακαθορίσουμε τους στόχους των σχέσεών μας με τη Λατινική Αμερική και να ε, τις τονίσουμε όπως χρειάζεται βάσει της λογικής που έχει περισχύσει τα τελευταία χρόνια εδώ. Ευχαριστώ. Έχουμε κάποιο χρόνο. Αρκετοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Να σας θυμίσω ότι είναι μια αρχική ακρόαση, θα συζητήσουμε μετά πολιτικά τα διάφορα ζητήματα. Ελπίζω διάφοροι να θέσουν θέματα στους εμπειρογνώμονες και ο καθένας θα έχει τη θέση του 1,5 λεπτό. Παρακαλώ σήμερα μόνο ερωτήσεις και η πολιτική συζήτηση θα διεξαχθεί ε, στα πλαίσια της προτάσης ψηφίσματος. ΕΛΚ. Ο κ. Σαλαφράγκα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ όλους τους ε, ομιλητές και τον εισηγητή μας, τον κύριο Λόπεθ. Η συζήτηση αυτή γίνεται υπό το φως ιδιαίτερων συνθηκών κάτω από τις οποίες βρίσκεται τόσο η Λιτινική Αμερική όσο και η Ευρώπη. Πριν από λίγο συζητήσαμε για τις εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες που μας έλεγε λίγο πολύ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, μα έχει αλλάξει. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και στη σχέση μας με την Λατινική Αμερική. Είδαμε τι γίνεται το κατακαιρμό των Άνδεων για τις σχέσεις με, τη... με τον Ειρηνικό των ΗΠΑ. Τα εξήγησε και ο κύριος Λόπες ότι μερικές φορές οι περιφέρειές μας ασχολούνται με τα δικά τους ζητήματα και ξεχνάμε τις σχέσεις μεταξύ μας. έγινε ο υπουργικό διάλογος στα πλαίσια του Ρίου. Ε, δεν φτάνουν όμως όλα αυτά. Ερχόμουν εδώ και διάβασα κάτι εδώ στον τρίτο όροφο που λέει ότι για να φτιάξει κανείς το μέλλον πρέπει να το δημιουργήσει. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Και νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει τις δυνατές και καλές σχέσεις. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα έπρεπε να κάνει μια δήλωση, τα ξέρετε πολύ καλά γιατί έχετε τεράστιο διπλωματικό παρελθόν, που να τονίζονται οι σχέσεις αυτές, οι περιφερειακές και οι παγκόσμιες, και να ενισχυθούν οι συμφωνίες τις οποίες θέλουμε να προσαρμόσουμε αυτή την εποχή εξαιτία των νέων καταστάσεων. Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η κυρία, με συγχωρείτε πολύ, η κυρία μισή λεπτό παρακαλώ. Μην ανησυχείτε πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα έχουν ήδη και από τον Χαμπί Λόπεθ αλλά και από τον συνάδελφο Σαλαφράγκα. Και όταν επαναλάβω αυτά που ακούσαμε από τους ομιλητές μας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και συγχαρητήρια σε όλους για την οργάνωση ακρόαση αυτής. Λοιπόν, θέλω όμως να είμαι και ρεαλίστρια. Κοιτάξτε την αίθουσα μαύρη τρύπα. Πάντα ίδιοι είμαστε εδώ, εδώ και 15 χρόνια. Εγώ έφυγα από το κοινοβούλιο για μερικά χρόνια, επανήλθα, την ίδια εικόνα όμως βλέπω. Εντάξει, υπάρχουν νέα κεφάλια που βλέπω, αλλά τι είμαστε, περισσότεροι Ισπανοί, κάποιοι λίγοι συνάδελφοι από άλλες χώρες που ενδιαφέρονται για τη Λατινική Αμερική. Σίγουρα μπορούμε να βασιστούμε στον συνάδελφο Χάμπι Λόπες, αλλά είναι κατάφορο ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είμαστε σε θέση να περάσουμε κάτι που για μας είναι προφανές, δηλαδή το πόσο σημαντικές είναι στέρες και ισχυρές σχέσεις Ευρώπης, Λατινικής Αμερικής. Τι είπαν οι συνάδελφοι, τι εργαλεία έχουμε, πώς προχωρούν τα πράγματα. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στον κόσμο ολόκληρο και αν μη τι άλλο, για λόγους ανάγκης, θα έπρεπε να δώσουμε νέα όθηση στην σχέση αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να επιταχύνουμε την όθηση αυτή. Η έκθεση Χάμπι Λόπετ, που θα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, ελπίζω να συνεισφέρει σε αυτό. Πάντως, σας διαβεβαιώ ότι δεν έχουμε πετύχει ακόμα τίποτα και χρειαζόμαστε και τη δικιά σας στήριξη και εννοείται ότι είμαστε στη διάθεσή σας. Ελπίζω να τα καταφέρουμε πριν να είναι πολύ αργά. Ο κύριο Τάνοκ, 1,5 λεπτό τώρα. η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, όπως είπατε και εσείς, επιτυχημένες εμπορικές ε, σχέσεις με ε, Χιλή, Κολομβία, Περού. Πώς μπορεί κανείς να επανεκκινήσει την ε, Συμφωνία Εμπορικών Συναλλαγών, Ελευθέρων Συναλλαγών με την Μερκοσούρ. Το μέγα πρόβλημα βεβαίως ήταν πάντοτε τα αγροτικά προϊόντα. Μήπως μπορείτε να Εξηγήστε πώς μπορεί να ξεπεραστεί το κόλλημα αυτό, διότι για μένα είναι σαφές ότι αυτό απέτρεψε την υπογραφή την τελευταία φορά. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λέφλερ είναι η Βρετανική έξοδος από την Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση. Brexit και οι συμφωνίες με τις οικονομίες της Καραϊβικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιτρέψει παράλληλες διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρετανικής κυβέρνησης και με τις χώρες αυτές όταν θα αρχίσουν ε, τους επόμενους μήνες, εκτός από τις διαπραγματεύσεις δηλαδή ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προωθήσει κυρίως την αγγλοσαξονική σφαίρα η ε, Βρετανική κυβέρνηση, δηλαδή με Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία, αλλά υπάρχουν και πολλές χώρες του ΑΚΕ οι οποίες θα θελήσουν να ε, συμφωνήσουν με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το άλλο τώρα είναι οι νέες σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής υπό τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση και με τον επαπειλούμενο τείχο του Μεξικού. Ιδίω βέβαια εάν η ναύτα η οποία τώρα επανεξετάζεται δεν υποστηριχθεί πλέον από την ε, Ουάσιγκτον. Βέμπερ, φιλελεύθερη, 1,5 λεπτό. Αρχίζω ευχαριστώντας πρώτα τον κύριο Λόπες που ανέλαβε την πρωτοβουλία για την οργάνωση της συναντήσεως. Ευχαριστώ όλες τις προσκεκλημένες που είναι πολύ σημαντικό βέβαια να τις ακούσουμε και να έχουμε επομένως πληροφορίες από πρώτο χέρι. Πολύ ευχαριστώ ακούω που λέτε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ ευχαριστώ άκουσμα για μένα. Ωστόσο, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε στρατηγική εταιρική σχέση και θεωρώ ότι προς τα εκεί πρέπει να κατευθυνθούμε, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις προκλήσεις που φέρνουν τα επόμενα χρόνια. Και εννοώ βεβαίω και την κλιματική αλλαγή, που αυτή θα επηρεάσει θέματα μετανάστευσης στο μέλλον. Βεβαίως και την ψηφιοποίηση, που θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και την παραγωγικότητα και την απασχόληση των ε, ανθρώπων καθώς και την κινητικότητα των ανθρώπων ε, στο πλαίσιο αυτό. Πέρα από το βάθεμα των συμφωνιών συνεργασίας, είμαι υπέρ αυτού και το υποστηρίζω, νομίζω όμως ότι χρειαζόμαστε ακόμη να προβλέψουμε κάπως το τι θα γίνει στο μέλλον και να κινηθούμε προς τις σωστές κατευθύνσεις. Και θέλω να πω στην αγαπητή μου φίλη Έλενα ότι εδώ ναι μεν είμαστε συνήθις ύποπτοι στην αίθουσα, η αλήθεια όμως είναι ότι υπάρχει ε, ενισχυμένη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Μάλιστα ευχαριστώ, επανέρχομαι στην ομάδα του Λαϊκού Κόμματος, ο κ. Τεγκράντης για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας, τον κύριο Λόπεθ και Ευχαριστώ πολύ όλους τους προσκεκλημένους μας που είναι τόσο ξέχουσες προσωπικότητες και λαμπροί. Σημειώνουμε λοιπόν τόσα είπανε. Και εγώ που είμαι σκιώδη εισηγητής για την έκθεση αυτή σημείωσα τόσα είπατε. Υπόθηκαν πράγματι πολλά σημαντικά εδώ. Είναι αλήθεια όπως είπε η Βέκα, ότι είναι μια στιγμή ευκαιρίας αλλά και προβληματισμού θα πρόσθετα εγώ, μετά από μία δεκαετία χρυσή για τη Λατινική Αμερική, το γεγονός ότι δεν υπάρχει οικουμενική προστασία είναι κάτι που οδηγεί σε προβλήματα. Είπατε ότι επανέρχεται η ανισότητα, άρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία και για την Ευρώπη να καλύψει ε, το κενό εκείνο το οποίο δεν κάλυψε ποτέ μέχρι τώρα. και ίσως οι διατλαντικές ε, σχέσεις που ήταν πάντα καλές τώρα είναι ακόμα πιο θετικές με τη Λατινική Αμερική. Η Ευρώπη θα πρέπει να φροντίσει να βρεθεί εκεί που πρέπει να καλύψει το κενό που υπάρχει και μερικές φορές εμείς είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Λοιπόν, πράγματι τα τελευταία δέκα χρόνια είχατε την χρυσή δεκαετία Τώρα τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύονται, γι' αυτό και εμείς πρέπει να φροντίσουμε, να καλύψουμε το κενό και να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Σοσιαλιτές, άσεις. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία της εκπονήσεως μιας εκθέσεως και της διοργανώσεως της ακροάσεως αυτής που διεξάγεται σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ζούμε ιδιαίτερες ε, στιγμές που έχουν συνέπειες για τις σχέσεις μας με τη Λατινική Αμερική. Υπήρξε μια φάση μεγάλης εφορίας και τώρα είμαστε σε μια φάση απογοήτευσης. Απογοήτευσης η οποία παράγει αντιδράσεις σε κάποιες χώρες και σε κάποιες περιφέρειες του κόσμου. Με αντιδράσεις οικονομικού προστατευτισμού που αρχίζει να διαφαίνεται και με απώλεια εμπιστοσύνης που παρατηρούμε ε, εν γέννη. Άρα η πολυμερής προσέγγιση ε, αμφισβητείται και πρέπει να επεξετάσουμε τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων περιοχών του κόσμου. Δυστυχώς η Ευρώπη δεν έχει ξεφύγει από αυτά τα αντανακλαστικά, τα προστατευτικά, του προστατευτισμού. Γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε επιτομέων που μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Πρέπει να επικεντρωθούμε επί της Λατινικής Αμερικής. Όπως αναφέρθηκε, μοιραζόμαστε κάποιες αξίες. Έχουμε τον ίδιο τρόπο προσέγγισης των μεγάλων διεθνών προβλημάτων. Άρα πρέπει να βασιστούμε περισσότερο στη σχέση αυτή μεταξύ Λατινικής Αμερικής και Ευρώπης και είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρώπη να στείλει αυτό το μήνυμα στις διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ δεν θα πρέπει η συνθήκη αυτή να παραμείνει παγωμένη όπως έγινε επί πολλά χρόνια. Για να κλείσουμε. Ραμύρες για το ΕΛΚ για 1,5 λεπτό. Ορίστε. Α, δεν κατάλαβα το όνομα μου, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη. Ευχαριστώ και εγώ, όπως και οι συνάδελφοι, τον εισηγητή πρώτα απ' όλα για την οργάνωση της συνάντησης αυτής και φυσικά και θέλω να ευχαριστήσω και τους ομιλητές και να ζητήσω συγγνώμη που άργησα να φτάσω. Όπως το πάνε η στιγμή αυτή είναι πολύ σημαντική. Εγώ επιστρέφω από το Μεξικό. Πήγα εκεί με την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις μας με το Μεξικό και υπήρχε και μέρος της ΣΥΝΤΑ. Η στιγμή είναι πολύ ιδιαίτερη. Πάντα έλεγα ότι η Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δίνει πάντα την προτεραιότητα στην ε, Λατινική Αμερική, αλλά ούτε και η Λατινική Αμερική δίνει προτεραιότητα στην Ευρώπη. Μεξικό, για παράδειγμα, πάντα θαύμαζε την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι βέβαια και δίπλα τους, αλλά ίσως πρέπει να αλλάξει αυτό. 80% βέβαια η οικονομία του Μεξικού εξαρτάται από τις Ηνωμένε Πολιτείες και όταν ξαφνικά εμφανίζεται ένας κύριος Τραμπ που τους λέει ότι θα φτιάξει το τείχος ή μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας Ναύτα, όλα αυτά βέβαια ακούγονται πολύ βία για τους Μεξικάνους, οι οποίοι είναι ευάλωτοι. Συνεπώς, ήρθε η στιγμή το Μεξικό να αποτελέσει για την Ευρώπη ένα σημαντικό εταίρο. Και η στιγμή αυτή μπορεί να βοηθήσει να υπάρξει προσέγγιση ανάμεσα στην Ευρώπη και ε, Μεξικό, Λατινική Αμερική κλπ. Είμαστε που επιζωνή χρονικά. Δυόμιση λεπτά ο κάθε εμπειρογνώμων για να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ζητώ συγγνώμη. Καμιά φορά οι πολιτικοί μακρηγορούν και στο τέλος υποφέρουμε από το χρόνο. Ακολουθήσουμε την σειρά. Ο κύριος Λέφλερ αν μπορεί να δώσει πρώτες απαντήσεις σε δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ για τα σχόλια, για τις ερωτήσεις. Τα σχόλια καταδεικνύουν σύγκληση όσον αφορά τη σημασία και την αξία της σχέσης αυτής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί. Ο κ. Τάνοκ ρώτησε για τις διαπραγματεύσεις Μερκοσούρ Πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα πια, να θυμηθούμε ότι η γεωργία παραμένει σημαντικός τομέας για τις χώρες Μερκοσούρ και για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όμως είναι πολύ μικρό κομμάτι των σχέσεών μας με το Μερκοσούρ και με τις διάφορες χώρες του Μερκοσούρ. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερο δυναμικό σχέσεις, οικονομικό, δυναμικό, πολιτικό και τεχνικό και θέλουμε να τα εκμεταλλευτούμε αυτά τα στοιχεία. Στην Καραϊβική, αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορεί να ξεκινήσει παράλληλε διαπραγματεύσει. Υποθέτουμε ότι όσο είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ενώση του Ηνωμένου Βασίλειου θα υποστηρίζει πιστά τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Η εμπορική πολιτική είναι κοινή πολιτική και ακρογωνίω λήθο των εξωτερικών μα σχέσεων. Όσον αφορά την αντικατάσταση τη ΝΑΦΤΑ, δεν αντικαθιστούμε την ναύτα, ελπίζουμε να εξακολουθεί να ισχύει η ναύτα. Δεν αντικαθιστούμε εμείς της ΕΠΑ στη Λατινική Αμερική, διότι από πλευρά επενδύσεων και εμπορίου είναι η πιο σημαντική Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λατινική Αμερική, με την εξαίρεση του Μεξικού λόγω των κοινωνικών σχέσεων. Αλλά δεν θα χτίσουμε τύχη σίγουρα, έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία κατεδαφίσεως τυχών παρά οικοδομήσεως αυτών. Μου τελειώνει ο χρόνος να τονίσω κάποια άλλα στοιχεία που αναφέρθηκαν. Επιστρέφοντας τα αρχικά μου λόγια. Έχει σημασία συνεργασία για την αλλαγή του κλίματος. Πολυμερός και έτσι δικές μας κοινωνίες. Στους τελευταίους μήνες κοιτάξτε τι έγινε στην Καραϊβική και στη Λατινική Αμερική. Καταστροφές λογοτυφώνων στην Κεντρική Αμερική και στην Καραϊβική. Ξηρασία στη Βραζιλία, πλημμύρες στο Περού Παρόμοια προβλήματα είχαμε σε κάποια μέρη της Ευρώπης. Αυτό είναι σαφέστατη ένδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, για τη συνδυσιμότητα, πριν από δύο χρόνια λάβαμε πρωτοβουλία να ξεκινήσουμε σχέση, ε, διασύνδεση με οπτικές ίνες μεταξύ Λατινικής Αμερικής και Ευρώπης προς όφελος των επιχειρήσεων, της έρευνας και των πολιτών. Τέλος, πολλά από αυτά που αναφέρθηκαν και πολλά από αυτά που είπατε και εσείς αξιότιμα μέλη και άλλα μέλη του πάνελ αφορούν αποτελεσματικότερη συνεργασία όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, δημιουργία ισχυροτέρων κοινωνιών, μοιράζοντας τα ωφέλη της παγκοσμιοποίησης και αντιμετωπίζοντας από κοινού τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρίνσπαν, ο κύριος Γκρίνσπαν. κυρία Γκρίνσπαν. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας, όλα πολύ ενδιαφέροντα. Συμφωνούμε. Αλλά θέλω να σας μεταφέρω κάποια μηνύματα έτσι, πολύ συγκεκριμένα. Πρώτον, οι ευκαιρίες που ανοίγουν κλείνουν κιόλα. Οπότε, υπενθυμίζω ότι η Κίνα τα τελευταία χρόνια, από το 2000 μέχρι το 2015, πολλαπλασίασε επί 22 το εμπόριό της με τη Λατινική Αμερική και αποτελεί μια πηγή χρηματοδότησης και μια πηγή επενδύσεων. Ο ειρηνικός θα εξακολουθεί να είναι σημαντικός, ε, δεν λέω, αλλά η Λατινική Αμερική δεν μπορεί να στοιχηματίζει μόνο στην Ασία. Πρώτες αγροτικά προϊόντα, υποδομές. Δεν μας φτάνει η Κίνα για την νεολαία μας και για το μέλλον της. Γι' αυτό λέω ότι έχει η Ευρώπη μία ευκαιρία. Μη μας διχάζετε ανάμεσα στη, στον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό. Εμείς θέλουμε να τα συμπεριλάβουμε και τα δύο. Είμαστε χώρες, Λατινική Αμερική, ανάμεσα σε δύο ωκεανούς. Και άρα πρέπει και με τις δύο πλευρές να συνεργαζόμαστε. Δεύτερον, χρειαζόμαστε συνεργασία, όπως είπε και η Πάολα, πιο οριζόντια πιο εγκάσια, πιο περιφερειακή, πιο θεματική. Μην μπαίνουμε σε διμερείς μόνο σχέσεις και θέματα. Χρειαζόμαστε πιο πολλά. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στην εκπαίδευση, στις επιστήμες, προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται όλες οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις, κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά γίνονται θεμελιώδους σημασία. Οπότε μην ε, χωρίζουμε την ε, περιοχή προσπαθώντας ε, στη μία να κάνουμε το ένα και στην άλλη χώρα το άλλο. Έπειτα έχουμε σημαντικά εργαλεία, τη Eurolat και τη διάσκεψη, που αποτελούν δύο μέσα πολύ σημαντικά πολιτικού διαλόγου και τα οποία φτιάχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Να τα προσέχουμε λοιπόν για να πετύχουμε τους στόχους πάνω στους οποίους όλοι συμφωνούμε για τις συμφωνίες και για τη συνεργασία και φυσικά το διάλογο μεταξύ των δύο περιοχών. Ευχαριστώ πολύ. And very keeping the time. Πολύ εντυπωσιακά τηρήσατε το χρόνο. Πολύ αποτελεσματική υπήρξατε. Τηρήσατε τα δύο μισή λεπτά. Έχετε εσείς το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κάτι το οποίο βγαίνει από τις παρεμβάσεις είναι η πρόκληση του να τα αποκραθούμε σωστά. Πώς να αποφύγουμε δηλαδή να βρεθούμε μέσα σε ένα κενό χρόνου όπου τελικά δεν ε, αλλάζει τίποτα. Όσον αφορά τις προκλήσεις και να τις αντιμετωπίσουμε έχουμε πολλά μέσα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ μας. Η σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική είναι ποιότητας. Αυτά που προσφέρει είναι ποιότητας. Και η επένδυση που κάνει η Ευρώπη στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική είναι επένδυση με κοινωνικές προδιαγραφές, οικολογικές προδιαγραφές, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει απαραίτητα <clears throat> από άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτό είναι το θετικό στις σχέσεις, έτσι όπως επίσης οι πολλές ε, ανταλλαγές που υπάρχουν σε επίπεδο θεσμικό, επιχειρήσεων, ε, πολιτών. Έπειτα, η επιτυχής ιστορία που έχουμε όσον αφορά την μετανάστευση από την ε, μία περιοχή στην άλλη και τούμπαλιν. Γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσει η αλληλοστήριξη. Αυτό που είπε ο κύριος Σαλαφράγκα τώρα, ότι πρέπει να φτιάξουμε το μέλλον. Η πρώτη επένδυση που πρέπει να κάνουμε και το πώς θα την κάνουμε είναι να δούμε πώς ε, αυτήν, την, ε, αυτό το δίλημα το αν θα είναι ε, σε διαφορετικό βαθμό ή ενιαία η σχέση αυτή. Πώς θα εξηγήσουμε σε ένα φοιτητή από τη Χιλή ότι δεν θα μπορέσει να συμμετέχει στο Ερασμός. Ενώ άλλοι ναι. Ένα μεγάλο πλονέκτημα της σχέσης αυτής είναι το ότι είναι θεσμική. Αλλά προσοχή, γιατί τελικά μπορεί να πνιγούμε στην γραφειοκρατία, κάτι το οποίο δεν θέλουν οι πολίτες. Να προσπαθήσουμε να βρούμε λοιπόν τρόπους να συμμετάσχουν στη σχέση αυτή όλες οι ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Ας δούμε αν και η τρίτη παρέμβαση θα τηρήσει τα 2,5 λεπτά. Όπω υπόθηκε ήδη, το θέμα αυτό των ευκαιριών είναι πολύ σημαντικό. Ότι δηλαδή η σημερινή πολιτική των ΗΠΑ μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την Ευρώπη στη σχέση της με τη Λατινική Αμερική. Κοιτάξτε, δεν είναι θετικό βέβαια οι Ηνωμένε μονομερός να υιοθετούν μια στάση προστατευτική κτλ. Είναι κάτι αποσταθεροποιητικό για όλους. Οπότε η συμμαχία της Ευρώπης με τη Λατινική Αμερική πρέπει να χρησιμεύσει για να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προχωρήσουν σε αυτό το δρόμο, γιατί οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σημαντικές έτσι κι Άρα να κάνουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να έρθουν στο δικό μας τρόπο σκέψης. Τώρα το θέμα θα πρέπει να υπάρχει διαβάθμιση όχι στις σχέσεις. Νομίζω ότι είναι ένας ε, μηχανισμός από τον οποίο υποφελούνται όλοι και η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική. Αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα. Μπορεί να τα βλέπουμε από διαφορετική οπτική γωνία, να έχουμε διαφορετική δυνατότητα αντιμετώπισης, αλλά ε, μας ε, βοηθάει η σχέση να βλέπουμε ε, μαζί προβλήματα τα οποία είναι παγκόσμια. Η παγκοσμιοποίηση ακριβώ μας κάνει να έχουμε τα ίδια προβλήματα τελικά μεταξύ μας. Ό,τι επηρεάζει τη, σημείο του κόσμου επηρεάζει και κάποιο άλλο. Η συνεργασία είναι επένδυση, είναι βοήθεια στο μέλλον, είναι δημόσιες δαπάνες που χρειάζονται και στη Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη αλλά φυσικά πρέπει να υπάρχει σωστή κατανομή, έτσι όπως γίνεται κάθε φορά με τις δαπάνες. Αυτό δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ε, ε, oh, Πήγατε, ε, ξεπεράσατε, σπάσατε τα ρεκόρ. Ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες που συνέβαλαν στις εργασίες μας. Ο εισηγητή και οι σκιώδει εισηγητέ έχουν πολύ καλέ πληροφορίε για να προχωρήσουν. Ευχαριστώ όλου που συμμετείχαν στην ακρόαση. Ολοκληρώνουμε για την ώρα τη συνεδρίασή μα και θα ξαναρχίσουμε στι 3 μετά το γεύμα. Και αφού συμμετάσχουμε στην επέτειο για τα 60 χρόνια τη συνθήκη τη Ρώμη, ευχαριστώ για την παρουσία σα. Τα λέμε αργότερα το απόγευμα. Γεια σα, καλή όρεξη.